Wprawdzie Πολύ σωστά ο κύριος Άγνιο μου υπενθυμίζει ότι είναι ώρα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Συμφωνείτε? Λέω κύριε Άγνιο, εσάς περίμενα να μου υπενθυμίσετε ότι είναι ώρα να αρχίσουμε, γιατί εσείς συνήθως ε, ε, μου επισημαίνεται ότι πρέπει να είμαστε ακριβείς και συνεπείς και να ξεκινάμε στην ώρα μας. Πέρασε όμως ακόμη και το ακαδημαϊκό τέταρτο και επειδή έχουμε ένα πανεπιστημιακού σεμιναρίου εδώ, σκέφτηκα σκόπιμο να αφήσω να κυλήσει το ακαδημαϊκό τέταρτο. Γιατί έχουμε πανεπιστημιακούς εδώ και είπα να σεβαστώ το δικό του ακαδημαϊκό τέταρτο και ταυτόχρονα περιμένω και τους ευρωβουλευτές για να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση. Ας αρχίσουμε όμως. Θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της δημόσιας αυτής ακρόασης και να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες αυτήν. Να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές για την παρουσία τους και να σας ε, ενημερώσω ότι ο πρώτος μας ομιλητής είναι ο κύριος Βιόλα που είναι ο διευθυντής ε, του ιδρύματο Edmund Mach ε, της, του Ερευνητικού και Κοινοτόμου Κέντρου της Ιταλίας. Δυστυχώς όμως ε, ασθενή και δεν μπόρεσε να έρθει. Ελπίζω σε μια μελλοντική δημοσιακρόση να μπορέσει να έρθει. Στόχος της σημερινής ε, δημόσιας ακρόασης είναι να εξοικειωθούν τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας με τα θέματα της βελτίωσης των φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός και να ε, ενθαρρυνθεί μια γενική συζήτηση για τις μελλοντικές προοπτικές της βελτίωσης ε, των φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινός μας στόχος είναι η εξασφάλιση του δυναμικού του φυτικού κλάδου και την αξιο... και η αξιοποίηση των ευκαιριών του, προκειμένου να προσαρμοστεί στις τοπικές ε, και περιφερειακές καθώς και ευρωπαϊκές ανάγκες στο μέλλον θα έχουμε δύο μέρη στην ακρόαση. Στο πρώτο τμήμα της θα επικεντρωθούμε σε επιστημονικές πληροφορίες για την σημερινή κατάσταση και τις προτεραιότητες της επιστήμης και της έρευνας στον τομέα αυτό και στο δεύτερο τμήμα θα ακούσουμε την γνώμη των ενδιαφερομένων. Μετά από, την μετά από το κάθε τμήμα της ακρόασης θα ακολουθήσει γύρω σε ερωταπαντήσεων. Όπως σας είπα, ο κύριος Ρομπέρτο Βιόλα δεν μπόρεσε να έρθει Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στο δεύτερο μας καλεσμένο, τον ε, κύριο Σλαβόμιρ Σόβα, που είναι επικεφαλής ε, του Εργαστηρίου Ελέγχου Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών ε, και του σημαντικότερου ερευνητικού Ινστιτούτου στην Πολωνία, το οποίο ασχολείται με τη βελτίωση των φυτών και τον εγκληματισμό. Έχει πολυκλαδικό προσανατολισμό το Ινστιτούτο αυτό και ασχολείται με τη βελτίωση των καλλιεργιών, τη βιοτεχνολογία, τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό του ιδιοπλάσματος. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον δόκτορα Σουαβόμιρ Σόβα, τον οποίο και ευχαριστώ που ήρθε και έχει ένα δεκάλεπτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ενημερώσω για τις νέες ε, τεχνικές βελτίωσεις των φυτών. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, δεν θα επικεντρωθώ στις τεχνικές πτυχές ε, των νέων τεχνικών βελτίωσης των φυτών, γιατί η πρόθεσή μου είναι να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το ρόλο της καινοτομίας στην αηφόρο γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγη υπομονή για να διορθώσουμε το σύστημα. Ωραία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως η γεωργία που θα είναι βιώσιμη από γεωργική, οικονομική και κοινωνική άποψη έχει θεμελιώδη σημασία για να συμβάλλει στην, στην εξάλληψη της φτώχειας και στην ε, επιστημιστική ασφάλεια. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος αγωγιάς τροφίμων. Γι' αυτό έχουμε ευθύνη να κατευθύνουμε και τις αλλαγές στις τρίτες χώρες, ε, που είναι οι χώρες που παράγουν για μας τα τρόφιμα. Εν ολίγης, ε, θα πρέπει να παράγουμε περισσότερο με λιγότερους φυσικούς πόρους και με διαφοροποίηση των καλλιεργειών μας. Κάτι που είναι δύσκολο λόγω και των κλιματικών αλλαγών και της υποβάθμισης των αρρώσιμων γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας ε, χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, ζανιοκτώνων. Και μια άλλη πολύ σημαντική πρόκληση είναι η μείωση των διαφορών των αποδόσεων εσοδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν τέτοιε διαφορέ, υπάρχει τέτοιο χάσμα μεταξύ των κρατών μελών εσοδίες. Και έχουμε διαφορές και μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, αλλά έχουμε κάποιους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. Για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε πρόσβαση στην καινοτομία. Και ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα αυτό είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή βιοοικονομία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η βελτίωση των φυτών είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια όλων των φυτών και για κάθε χρήση, όχι μόνο για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών. Ο γεωργικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία μια βιοοικονομία που στηρίζεται στη γνώση για να αντιμετωπιστούν ε, οι προκλήσει τη επιστημική ασφάλεια, ε, του μετριασμού των κλιματικών αλλαγών και τη εξασφάλιση μια αηφόρου γεωργίας. Υπάρχουν πολλέ τεχνικέ βελτίωσει των φυτών. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για νουκλεάσες δακτύλου ψευδορύρου, ε, αναστροφές, διάφορες ε, ε, τεχνικές βελτίωσης ε, προχωρούν και προοδεύουν ραγδαία και θα έχουμε όλο και περισσότερες. Έχουμε ένα κατάλογο εδώ με τις νέες τεχνικές βελτίωσεις. Δεν είναι όμως όλες καινούριες. Για παράδειγμα, η, μεταμόσχευση, η μεταμόσχευση, η cisgenesis, intragenesis είναι γνωστές όπως και η έχει εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, ε, έχουμε την ομογονιδιακή τέτοια γενετική επεξεργασία που είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να αποκτήσουμε πιο ανθεκτικά φυτά. Για παράδειγμα, το παράσιτο φυτοφθόρα infestans, που είναι το πιο σημαντικό παθογόνο της πατάτας και προκαλεί τον περονόσπορο. Τα περισσότερα μικητοκτόνα που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες χώρες χρησιμοποιούνται ακριβώ για να εξολοθερθεί αυτό ο ομίκητο που προκαλεί τον περονόσπορο. Υπάρχουν όμω και κάποιε τεχνικέ διόρθωση του γονιδιώματο. Γίνονται μικρέ αλλαγέ στο γονιδίωμα των οργανισμών. Πρόκειται όμω και για αλλαγέ που μπορούν να λάβουν χώρα και με φυσιολογικό τρόπο. Οπότε αντί να περιμένουμε τι τέτοιε αλλαγέ από τη φύση με μια φυσιολογική διαδικασία, κάτι που είναι πολύ χρονοβόρα, ή να, αντί να χρησιμοποιούμε χημικέ μεθόδου ή ακτινοβολία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα, ένα πιο στοχευμένο και ακριβή τρόπο. Μία μικρή αλλαγή στην αλληλουχία του DNA σε ένα νουκλεότυπο μπορεί να δημιουργήσει τεράστια πλεονεκτήματα για τους βελτιωτές και να εξασφαλίσει, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των φυτών στα φυτοφάρμακα και στο στρες. Με βάση την οδηγία του 2001-18 αναφέρεται ότι η γενετικός τροποποιημένος οργανισμός είναι ένας οργανισμός που το γενετικό του υλικό έχει τροποποιηθεί με τρόπο που περιλαμβάνει και τον ανασυνδυασμό του νεκλινικού οξέως. Αυτός είναι παλιός ε, ορισμός, προ 25 ετίας ε, και δεν έχει επικαιροποιηθεί. Ε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί είναι οργανισμοί με νέες ε, με νέους γονιδιακούς συνδυασμούς που ξεπερνούν τα φυσικά όρια του, της σύζευξης ή του ανασυνδυασμού. Τώρα, αν κοιτάξουμε εκ του στην οδηγία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σειρά τεχνικών όπως είναι ανασυνδυασμός νουκλινικού οξέως, άμεση ε, εισαγωγή ή κάποιες τεχνικές που δεν οδηγούν σε μετασχηματισμό των γονιδίων, για φυσιολογικές διαδικασίες ε, μεταμόρφωσης μετασχηματισμού. Επίσης υπάρχει τεχνικές που ε, θεωρούνται ως γενετική τροποποίηση, αλλά εξαιρούνται από την οδηγία, όπως είναι η μεταλλαξογένεση, που είναι βασικό στοιχείο της φυσιολογικής διαδικασίας εξέλιξης. Με βάση λοιπόν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ένα προϊόν θεωρείται γενετικώς τροποποιημένο με βάση την διαδικασία με την οποία έχει παραχθεί και το προϊόν. Ο... Η Οδηγία 1829 του 2003 απαιτεί επισήμανση για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές και μάλιστα ο τρόπος ε, ταυτοποίησης, ε, εντοπισμού και ποσοτικοποίησης είναι τμήμα της διαδικασίας επισήμανσης ε, των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Βέβαια, ο εντοπισμός είναι γνωστός και εύκολος και χωρίς προηγούμενη γνώση της αλλαγής. Είναι εύκολο μερικές φορές να εντοπίσουμε, αλλά όχι και να ταυτοποιήσουμε την πηγή της αλλαγής γιατί αυτή η αλλαγή συμβαίνει με φυσιολογικό τρόπο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σαφέ, εναρμονισμένο σύστημα που θα εξασφαλίσει το εμπόριο γεωργικών προϊόντων σε προσιτέ τιμέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και ασφάλεια δικαίου για τι επιχειρήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πολιτικές με στόχο να προωθήσουν την καινοτομία στην γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων. Η καινοτομία όμως ε, δεν ε, είναι κάτι περιορισμένο. Φτάνει στους χρήστες, στους προμηθευτές, στους καταναλωτές, ξεπερνά τα σύνορα. Γι' αυτό και θα πρέπει να κατασκευάσουμε γέφυρες μεταξύ της έρευνας, της τεχνολογίας και των ενδιαφερομένων, των παραγωγών, των γεωργών, του κλάδου και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έτσι, η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία θα προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την αηφόρο ανάπτυξη. Αυτέ βέβαια είναι προσωπικέ μου απόψει. Πάντως πιστεύω ακράδαντα ότι οι νέες τεχνικές βελτίωσεις ε, δημιουργούν τεράστιε ευκαιρίε και για τι ε, βιολογικέ αγορέ, Γιατί βιολογική, τα βιολογικά τρόφιμα αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο και η οργανική παραγωγή θα παίξει μεγάλο ρόλο στην επιστημιστική ασφάλεια, γιατί σέβεται τον κύκλο ζωή και το περιβάλλον και έχει περιορισμένη χρήση και φυτοφαρμάκων και λοιπασμάτων. Και έχουμε όλο και μεγαλύτερη ζήτηση ε, ποικιλιών καλλιεργιών που θα αντέχουν στους επιβλαβείς οργανισμούς, στις αρρώστιες και στα βιωτικά στρες. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε την πρωτοπόρα θέση που έχουμε σε θέματα καινοτομία και έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στη γεωργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε γι' αυτό ασφάλεια δικαίου. Οι Ευρωπαίοι βελτιωτέ θέλουν να χρησιμοποιήσουν νέε τεχνικέ βελτίωσει, γιατί αυξάνουν την ταχύτητα και είναι και πολύ πιο ακριβεί οι παρεμβάσει. Και παρόλο που εκπίπτουν οι νέε τεχνικέ βελτίωσει από την νομοθεσία για τις γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού και γίνεται περιπτωσιολογικά η αξιολόγησή του, σίγουρα θα ευνοήσουν όλους μας. Ε, θα έχουμε, οι γεωργοί θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερες ποικιλίε. Αλλά και οι εταιρείε ε, θα μείνουν ανταγωνιστικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σπόρων και εξαγωγές σπόρων. Αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα υποφεληθούν από ασφαλέστερα τρόφιμα και καθαρότερο περιβάλλον. Επίσης, έρευνα και τεχνολογία νέων τεχνικών θα πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και οι αρμόδιοι και ενδιαφερόμενοι καλούν την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να υποβάλει σε προτάσεις. Και πριν από δύο εβδομάδες ε, το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας έγραψε ότι το CRISPR-Cas9, άρα επιδόψεις, το μετάλλαγμα αυτό που δεν περιέχει πια Cas9 ε, και στοχευμένα γονίδια RNA δεν θεωρείται ότι εμπίπτει στην νομοθεσία για, τα, για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Και έχουμε και μια καρικατούρα που λέει ε, μάλλον σας ε, ε, ανέβασα πολύ τις προσδοκίες φαίνεται ότι κάποιος έβαλε ένα φως στη μέση του τούνελ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε ιδιαίτερως που τηρήσατε και το χρόνο αγόρευσης. Θα περάσουμε στον επόμενό μας ομιλητή, τον καλεσμένο μας. Ε, προηγουμένως όμως θα καλωσορίσω μια ομάδα νέων ε, γεωργών από τη Γερμανία. Τους καλωσορίζουμε θερμά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που παρακολουθούν αυτή τη δημόσια ακρόαση. Πρόκειται για καλεσμένους του Νόρμπερτ Λίντς. Δεύτερη ομάδα από τη Γερμανία. Καλωσορίζω και εσάς. Έχουμε δύο ομάδες επισκεπτών δηλαδή από τη Γερμανία. Σας εύχομαι καλή διαμονή στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μας καλεσμένο, στον καθηγητή Ρίτσαρντ Βίσερ, που είναι ε, επικεφαλής του τμήματος βελτίωση των φυτών ε, στο Wageningen στις κατοχώρες θα μας παρουσιάσει την, τις τεχνικές ε, βελτίωσης των φυτών κυρίως στην πρωτογενή παραγωγή. Ο κύριος Βίσερ είναι εμπειρογνώμονα σε θέματα βελτίωση φυτών, μέλο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου στο Πανεπιστήμιο του Βάγκενιγκεν και έχει συντονίσει πολλά διεθνή προγράμματα στον τομέα αυτό. Είναι επικεφαλή και πρόεδρο πολλών διεθνών επιτροπών που αφορούν τη βελτίωση των φυτών, την πατάτα, βιοπληροφορική στη βελτίωση των φυτών και έχει δημοσιεύσει πάνω από 400 ε, κείμενα που έχουν γίνει σημεία αναφοράς για τον κλάδο. Σας ευχαριστώ. Ε, που ήρθατε κύριε καθηγητά και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά έρχομαι να ομιλήσω ενώπιόν σας και να συζητήσουμε πτυχές των νέων τεχνολογιών για την βελτίωση των φυτών. Αυτό που θα ήθελα να πράξω είναι να τονίσω όπως ο γειτονάς μου ότι οι τεχνικές βελτιώσεις είναι νέο πράγμα, αλλά αύριο θα είναι παραδοσιακό και μεθαύριο θα είναι ίσως και απειχιωμένες. Υπάρχει λοιπόν ε, η διαρκής ανάπτυξη των τεχνολογιών και πολλές από αυτές τις τεχνικές που ίσως είναι νέες για κάποιο είδος ε, μπορεί να είναι πια παλιές σε κάποιο άλλο είδος. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε διαρκώς υπόψη μας. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε με αρκετή ασφάλεια ότι οι νέες ε, τεχνολογίες αυτές είναι ένα συνηθισμένο πλέον ε, τμήμα αυτών των βελτιώσεων των φυτών. Πολλές από τις τεχνικές αυτές των τελευταίων πέντε ετών ας πούμε ε, επίσης, ε, δική μου γνώμη βέβαια είναι αυτή, είναι και καθιερωμένες πλέον για την αντιμετώπιση παλιών προβλημάτων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, λόγω της έλλειψης ξεκάθαρου ορισμού για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή όχι τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ότι αυτές οι νέες τεχνικές που έρχονται είναι ισχυρές μέθοδοι για να επιτύχουμε αυτό το precision breeding, την ε, ακριβή βελτίωση δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε δύο γονείς, τους διασταυρώνουμε και μετά καταλήγουμε σε ένα αριθμό νέων φυτών. Ο τρόπος για να βελτιωθεί και να γίνει πιο αποδοτική η ε, προσπάθεια αυτή και να ε, επιταχυνθεί ο κύκλος είναι αυτό που απασχολεί τώρα τι τεχνικές και ιδίω για εσοδίες που δεν είναι self-pollinating, δηλαδή δεν αυτοεπικονιάζονται όπως για παράδειγμα μήλα, μπανάνες και διάφορα άλλα. Εκεί οι τεχνικές αυτές είναι πολύ αποδοτικές και σημαντικές για την επίτευξη καλύτερων ποικιλιών. Ο γειτονά μου μίλησε για αυτές τις νέες τεχνικές και βέβαια η ε, λίστα μεγαλώνει διαρκώς. Επιτρέψτε μου τώρα να σας δείξω με ένα παράδειγμα την πατάτα και τον πελονόσφορο τι μπορεί να κάνει η πρακτική της cisgenesis, η διαδικασία cisgenesis για την πατάτα. Η πατάτα όπως θα γνωρίζετε είναι η τρίτη μεγαλύτερη εσοδεία στον κόσμο, είναι παγκόσμιας ε, σημασίας και ε, ούτως ή άλλως παράγεται και παγκοσμίως και πάρα πολύ σημαντική και για το μέλλον έτσι ώστε να ε, υπάρχει παρκή ε, τροφή για τον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια πολλά προβλήματα. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι αυτή, αυτός ο περονόσπορος, ιδίως σε χώρες που έχουν κάπως ψυχρότερα κλίματα και ε, επαρκή βροχόπτωση. Εκεί η νόσος αυτή μπορεί μέσα σε μια-δύο εβδομάδες να καταστρέψει ολόκληρη την εισοδεία. Βλέπετε εδώ τον παράγοντα, δηλαδή τον επιβλαβή οργανισμό που ε, ονομάζεται στα λατινικά Phytophthora infestans και προκαλεί τον περονόσφορο. Και από τη στιγμή που θα πληγεί το φυτό δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα και θα καταστραφεί ολόκληρη η παραγωγή. Ούτως ή άλλως και θα πρέπει ε, να καταστραφούν διότι αλλιώς θα σαπίσουν και στις αποθήκες. Το ε, περιβαλλοντικό κόστος για τις κοινωνίες μας του Περονόσπορου είναι πραγματικά τεράστιο. Βλέπετε εδώ παράδειγμα προ 15 ετία, Ωστόσο τα νούμερα είναι συγκρίσιμα σήμερα. Βλέπετε ότι οι ε, Ολλανδοί γεωργοί έκαναν ε, τουλάχιστον 12 με 15 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο. Ε, βλέπετε και τον αριθμό χιλιάδων τόνων που χρησιμοποιούσαν ε, των ε, ουσιών και το κόστος για το συγκεκριμένο εκείνο χρόνο ήταν περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Εάν υπολογίσει κανείς την ποσότητα της πατάτας που ε, σε ολόκληρο τον κόσμο είναι βεβαίω τη τάξη των δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα κάτι πρέπει να γίνει για αυτή την ε, νόσο, για την καταπληκτική τη νόσου. εμείς. λαμβάνουμε γονιδίωμα από άγρια φυτά που είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτικά ορισμένα άγρια είδη σε, αυτόν, ε, σε αυτό το παράσιτο. Και αυτό που κάνουν είναι ότι μετακινούν μεταξύ των πληθυσμών τους τον αριθμό των ε, ε, ανθεκτικών γονιδίων. Δηλαδή η ασθένεια μπορεί να σκοτώσει ορισμένους γονιδιότυπους αλλά κάποιοι θα παραμείνουν ζωντανοί και έτσι διατηρείται ο πληθυσμός του είδους. Εάν κάνει κανείς τώρα τη διασταύρωση θα, θα δείτε ότι έχετε μητέρα, πατέρα και τα μισά γονιδιώματα της μητέρας και τα μισά γονίδια του πατέρα μεταφέρονται τελικά. Άρα δηλαδή όχι μόνο το γονίδιο της αντίστασης, της ανθεκτικότητας δηλαδή, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά μεταφέρονται με τα γονίδια από τα δύο ε, γονικά φυτά. Ένας από τους προκατόχους μου, ο καθηγητής ΕΜΣ, άρχισε ήδη από το 1950 την προσπάθεια διασταύρωσης ορισμένων από αυτά τα ανθεκτικά γονίδια, να τα μεταφέρει δηλαδή στην καλλιεργούμενη πατάτα. Η διαδικασία πήρε περίπου 45 χρόνια μέχρι ότου φτάσουμε σε δύο ποικιλίε την πιόνικα... Υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα με τη διαφάνεια. Τη βλέπετε πάνω-πάνω στη διαφάνεια αυτή. Και ήδη μετά από μία τριετία από την ε, χρήση της βρήκαμε ε, τα πρώτα εκείνα γονίδια τα οποία μπόρεσαν να ανακόψουν την ε, επέκταση της ε, ασθένειας. Είδατε 45 χρόνια μέχρι να γίνει αυτό το σημαντικό βήμα επιτυχίας. Αυτό βέβαια δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης ούτε και είναι δυνατό να είναι βιώσιμος. Από την άλλη μεριά αν χρησιμοποιήσετε γενετική τροποποίηση ή την cisgenesis, introgenesis ή intermutation breeding, αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την ποικιλία που διαθέτετε και να αλλάξετε μοναχά το γονίδιο εκείνο το οποίο σας ενδιαφέρει. Το κάνουμε αυτό με την διαδικασία της Genesis και με τον τρόπο αυτό εντοπίζετε το γονίδιο από ένα διασταυρώσιμο είδος, το παίρνει το γονίδιο όπως είναι και το βάζετε μέσα σε μια υφιστάμενη ποικιλία. Και αυτό που αποκτάτε εν τέλει, μέσα σε τρία χρόνια δηλαδή, είναι ότι μπορείτε να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα με μια μεγάλη διαφορά που είναι ότι η ελίτ ποικιλία είτε όπως και, ε, ε, όπως και να ονομάζεται ε, είναι γνωστή η ποικιλία αυτή και στη βιομηχανία και στους γεωργούς εξακολουθεί να υπάρχει αλλά περιλαμβάνει τώρα και κάποια ανθεκτικά γονίδια κατά της ασθένειας. Πολύ χρήσιμος τρόπος για να, για να εξασφαλιστεί η διατήρηση των ποικιλιών ελίτ. Το κάναμε αυτό την τελευταία δεκαετία. Και βλέπετε στη διαφάνεια που σας δείχνω τώρα μερικούς από τους κύκλους που κάναμε από το 2010 έχουμε κάνει μάλιστα πολλά επιτόπου στα χωράφια δηλαδή πειράματα, βλέπετε φωτογραφίες από τα πειράματα αυτά, βλέπετε χωρίς ψεκασμούς που κατάφερε το φυτό να ε, αντισταθεί στον περονόσπο. Επαναλαμβάνω, χωρίς ψεκασμούς. Δεν λέω ότι μπορούμε να εγκαταλείψουμε πολύ του ψεκασμού, μπορούμε όμω να του περιορίσουμε σημαντικά. Αυτό λέω. Και να εφαρμόζουμε ψεκασμού μόνο όταν δούμε ότι κάποια τμήματα τη φυτοφθόρα καταφέρνουν να ξεπεράσουν την αντίσταση των ε, ε, γονιδίων αντίσταση. Στην αριστερή πλευρά, για σας τώρα βλέπετε όλο και περισσότερα γονίδια να προστίθεται, βλέπετε ανάλογα με το κάθε παρτέρι και όταν έχετε πιο ανθεκτικά γονίδια βλέπετε τι ωραία που είναι τα παρτέρια αυτά και δεν υπάρχει απολύτως καμία ε, καταστροφή από την φυτοφθόρα. Και στη δεξιά πλευρά βέβαια είναι ψεκασμένα και εκεί διατηρείται βέβαια η εισόδια όπως έχει. Τα αποτελέσματα λοιπόν για την ώρα είναι ότι καταφέραμε να ε, μεταμορφώσουμε, ε, να μεταλλάξουμε δηλαδή 8 ποικιλίε πατάτας. Έχουμε 6 χρόνια τώρα ε, πειράματα επιτόπου στους αγρούς στην Ολλανδία και 2 χρόνια στο Βέλγιο και είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Όπως είπε εδώ ο γείτονά μου εκ δεξιών, πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε πιο βιώσιμες σοδιές με λιγότερη χρήση ε, και αυτό επομένως θα είναι μια πολύ χρήσιμη εξέλιξη σε, χρήση, σε συνδυασμό με όλες τις άλλες τεχνικές που διαθέτουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω με τη διαδικασία cisgenesis αλλά και με τις άλλες ε, ε, τεχνικές μετάλλαξης για διασταυρούμενες εσοδίες που Χρειάζεται βέβαια να μειωθεί ο χρόνος γιατί μπορούμε να μειώσουμε τα προηγούμενα 10 με 20 χρόνια να τα περιορίσουμε σε 5 και επομένως η προσπάθεια αυτή είναι πάρα πολύ αποδοτικότερη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Όντως, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων. Παρακαλώ. Ποιος θέλει το λόγο, κύριος Άγνιου. Σας ακούμε κύριε Άγνιου. Ήρθα μπροστά και κάθισα στη θέση κάποιου αλλού για να είμαι πιο κοντά στην παρουσίαση, για να σας ενοχλώ. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο κύριος ε, Βίσε. Δύο-τρία πράγματα έχω να ρωτήσω. Αυτά που μόλις μας περιγράψατε για τον περονόσπορο της πατάτας, αυτό είναι γονιδιακά ε, τροποποιημένο, μεταλλαγμένο ή... ή νέο τρόφιμο. Γιατί αν είναι GM τότε υπάρχει μεγάλη αντίσταση ε, από τον κόσμο. Αλλά αν δεν είναι GM ε, τότε μπορεί να περάσει αυτό. Ε, είπατε κάπου για ένα κόκκινο γονίδιο. Είναι το γονίδιο το οποίο έχει αντίσταση. Αλλά αναφέρατε και τρία άλλα κίτρινα γονίδια από την πλευρά του δωρητή. Δεν, δεν κατάλαβα γιατί ε, τα βάλατε και αυτά. Ε, απλά, ξέρετε, είναι δύσκολο να καταλάβουμε όλα τα επιστημονικά στοιχεία. Επίσης, ε, στις ε, καλλιέργειες έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Το ένα από τα δύο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ε, τεχνικές μετάλλαξες. Ε, το black grass που βρίσκουμε στα δημητριακά. Ε, δυστυχώς όμως η τεχνική αντιμετώπιση είναι ε, GM και το ότι δεν τη χρησιμοποιούμε κοστίζει τεράστια ποσά σε φυτοφάρμακα στη βιομηχανία και συχνά αποτυγχάνει τελικά θα μπορούσαν ε, οι νέες μέθοδοι που προτείνεται να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα του ε, black grass ε, ή πρέπει να είναι γονιδιακά μεταλλαγμένα σε όλες τις περιπτώσεις οι τρόποι αντιμετώπισης αυτού. Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά το αν είναι GM ή όχι. Ναι, σύμφωνα με τον ορισμό η διαδικασία της Genesis είναι GM αλλά είναι γενετικό τροποιημένη. Αλλά μετά από πολλές έρευνες έχουμε αντιληφθεί ότι το ευρύτερο κοινό βλέπει πολύ πιο θετικά την cisgenesis σε σχέση με την transgenesis. Έτσι ονομάζεται η άλλη μέθοδος. Αλλά ναι, είναι ε, μέθοδος γενετικής τροποποίησης. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τη μεταφορά περισσότερων γονιδίων. Ουσιαστικά εδώ γίνεται ουσιαστικά μια κανονική διασταύρωση και ουσιαστικά τα μισά γονίδια μεταφέρονται μόνο. Όχι μόνο δηλαδή το γονίδιο που μας ενδιαφέρει, το γονίδιο αντίσταση, αλλά και άλλα πράγματα. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στη βελτίωση των φυτών είναι να ξεφορτωθούμε όλα τα υπόλοιπα γονίδια. Γιατί δεν τα επιθυμούμε. Και εκεί αυτή είναι η αρνητική πτυχή ουσιαστικά. Αυτό τι σημαίνει ότι αν έχουμε μια τεχνική συσγένεσης, transgenesis ή νέας βελτίωσης, τότε ασχολούμαστε μόνο με το γονίδιο που μας ενδιαφέρει. Αυτό θέλουμε να βάλουμε στο φυτό. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει με την τρανσένεση και τη συστσέρεση. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά από τι νέε τεχνικέ βελτιώσει ξέρουμε ακριβώ τι κάνουμε. Οπότε είναι πιο ακριβή. Και τέλο, η τρίτη σα ερώτηση όσον αφορά το black grass ε, στα δημητριακά. Δεν γνωρίζω την ασθένεια που αναφέρεται. Ε, λοιπόν, το black grass ε, είναι ένα, ένα ζυζάνιο, όχι, δεν είναι ασθένεια. Ε, ονομάζεται αγρίο, ε, αλοπέκουρο ομοιόρο στα ελληνικά. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μετάλλαξη, βελτίωση μέσω μετάλλαξη. Ε, ίσως θα μπορούσε να βελτιώσει κανεί την αντοχή των Δημητριακών σε σχέση με το Ζιζάνιο. Äh, äh, Αυτές οι ε, τεχνικές θα πρέπει και να επισημαίνονται για να είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για φυσιολογικές διαδικασίες βελτίωσης. Βέβαια είναι και κρίσιμο το θέμα. Μου θυμίζει λίγο αυτά τα οποία εξηγήσατε εσείς οι δυο δηλαδή, ότι η, αυτό, που έχει αρχίσει η βιομηχανία γενετικών μεταλλάξεων ότι το μόνο που ενδιαφερόταν μας τα έλεγε αυτά πριν από 20 χρόνια ήταν να αυξήσει την ανθεκτικότητα των φυτών αλλά δεν πιστεύετε ότι είναι το ίδιο επικίνδυνο να πάμε τώρα σε τεχνικές βελτίωσεις που υποτίθεται ότι θα αποδώσουν τα ίδια που έλεγε τότε η βιομηχανία μετάλλαξης και που τελικά δεν απέδωσαν. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που ε, θα γίνει είναι να χάσουμε ποικιλία δηλαδή ε, βιοπικιλία, να χάσουμε ενδεχομένω ποικιλίε φυτών που ε, είναι ανθεκτικές και τελικά να μειωθεί το δυναμικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες. Και ένα πράγμα δεν κατανόησα πολύ καλά. Είπατε ότι όλα αυτά θα ενισχύσουν τη βιολογική γεωργία. Ε, sorry θα πω εγώ, όλη η βιολογική γεωργία αντιμετωπίζουν με μεγάλη επιφύλαξη όλες αυτές τις τεχνικές. Τα ίδια ακούγαμε όπως σας είπα και για τις τεχνικές μετάλλαξης προοικοσαετίας. Μας είχαν πει από τότε ότι άμα χρησιμοποιείς τεχνικές αυτές δεν θα χρειάζεται να ψεκάζετε. Τα είδαμε, δεν απέδωσαν τίποτα αυτά. Δεν είναι καθόλου πράγματα αυτά για τη βιολογική γεωργία και ούτε να τα βάζετε για διαφήμιση. Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά που είπε ο Χόισλινγκ, όντως πράγματι μετά από πολλές δεκαετίες δεν έχουμε προχωρήσει σε ό,τι αφορά τις τεχνικές ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Έχουμε στην ε, πατρίδα μου, το, ε, τη Ρόλο δηλαδή, πολλές καλλιέργειες αμπελιών κλπ. Και βλέπουμε ότι στην ουσία σημειωτών κάνουμε ακόμη και η μοναδική πραγματική ε, δυνατότητα που έχουμε για ίσως είναι χρήσιμες για ορισμένες ε, παραγωγές όπως, όπως εξήγησατε της πατάτας ίσως εκεί να είναι δυνατό να γίνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την μείωση των, ε, της χρήσης ανιοκτώνων. Φέρατε το παράδειγμα της διαδικασίας της Genesis για την πατάτα. Γνωρίζετε στην Ευρώπη πόσα φυτά ή πόσες καλλιέργειες υπάρχουν όπου έχει χρησιμοποιηθεί η πόσε καλλιεργειες υπαρχουν οπου εχει συγγένεσης. Τα επόμενα χρόνια πόσα φυτά θα μπουν στη διαδικασία της αναγνώρισης. Είναι σημαντικό το ερώτημα αυτό για να ορίσουμε και εμείς την τοποθέτησή μας. Όπως είπε και ο κύριος Σόβα, αρκεί να δούμε την πορεία της ε, γενετικής μετάλλαξης τα τελευταία 20 χρόνια, για να έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση μετά από τα σχόλια που ακούσαμε εδώ στην Επιτροπή. Μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πιστεύω ότι οι τεχνικές βελτίωσεις, οι νέες τεχνικές βελτίωσεις μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση. Δεν υπάρχει φυσικά τέλεια ε, λύση, δεν είναι πανάκια, είναι σε βελτιωτικές τεχνικές. Πιστεύω ότι ένας συνδυασμός με τη βιολογική διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών και ίσως και μαζί με τις νέες τεχνικές βελτίωσης και τα νέα χημικά, ένας συνδυασμός όλων αυτών θα μπορούσε να είναι η λύση. Τι πιστεύετε εσείς? Η κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, αυτές οι νέες τεχνικές βελτίωσεις που μας αναφέρατε επηρεάζονται από τον ορισμό των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, αν κατάλαβα καλά. Ποια είναι η δική σας πρόταση, τι αλλαγές προτείνετε ώστε αυτές οι νέες τεχνικές βελτίωσεις ε, να μην περιλαμβάνονται στον ορισμό για τα γενετικά τροποποιημένα. Και ο κύριος Μπούντα είναι ο τελευταίος σε αυτό το γύρο. Σας ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο καλεσμένους μας για τις παρουσιάσεις που μας έκαναν και να τους συγχαρώ για το έργο τους. Γιατί χωρίς τέτοιες προσπάθειες ε, δεν θα μπορούσαμε να προοδεύσουμε. Χρειαζόμαστε έρευνα, χρειαζόμαστε νέες τεχνικές. Οι αγρότες μας έχουν ανάγκη νέες τεχνικές. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, χρειάζεται επισήμανση των προϊόντων που προκύπτουν με τη χρήση τέτοιων τεχνικών βελτίωσης των φυτών. Στις δικές σας λοιπόν εκτιμήσεις και αξιολογήσεις περιλαμβάνονται κάποιες μελέτες για τη χρήση των φυτοφαρμάκων και τις τεχνικές μετάλλαξης και ποια είναι τα ωφέλη που προκύπτουν από τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα σε ό,τι αφορά την περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, για παράδειγμα. Και τι γίνεται για τους καταναλωτές. Είναι καλύτερο για τους καταναλωτές ε, να καταναλώνουν μεταλλαγμένα τρόφιμα ή τρόφιμα που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Δεν βλέπω άλλον κανένα να αναζητάει το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο τώρα στου δύο εμπειρογνώμονέ μα για να σχολιάσουν και να απαντήσουν. Συνονεθείτε μεταξύ σας ποιος θα είναι ο πρώτος. Okay. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και ζητώ συγγνώμη που άρχισα να απαντάω αμέσως μετά από το πρώτο άτομο που έβαλε ερωτήσεις. Λοιπόν, ως βέλτιο της ε, φυτών Θέλω να χρησιμοποιώ τι ε, πιο διαθέσιμε τεχνικέ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν λέω λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο τη γενετική μετάλλαξη. Λέω να χρησιμοποιούμε τι καλύτερε υπάρχουσε τεχνικέ, διαθέσιμε τεχνικέ, για να επιτυγχάνουμε τι καλύτερε καλλιέργειε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, χωρί να χρησιμοποιούμε υπερβολική ποσότητα φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών, ε, επιβαρύνοντα έτσι το περιβάλλον. Ε, είναι σίγουρα λιγότερο ασφαλέ από ό,τι θα θέλαμε. Επίσης ακούσαμε κάποια σχόλια για τις βιολογικές καλλιέργειες, ε, τις υποσχέσεις, την ε, παρακμή των ε, ποικιλιών. Ναι, αυτά αναφέρονται πάντα. Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε μια μελέτη για την παρακμή της ποικιλία των καλλιεργειών. Ναι, ο αριθμός μεν έχει μειωθεί. αλλά από τη δεκαετία του 70 πολλές καλλιέργειες βελτιώνονται όσον αφορά την ε, ποικιλία τους διότι χρησιμοποιήθηκαν πολλά είδη σε διασταύρωση μαζί τους για να βελτιωθεί η αντίσταση. Σίγουρα η πρόοδο στη βελτίωση των φυτών δεν υπήρξε τόσο ικανοποιητική, σίγουρα όχι σε όλε τι καλλιέργειε, γιατί αν δείτε το ζαχαρότευτλο για παράδειγμα θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στην αντίσταση λόγω των ε, νέων τεχνικών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι ένα πολύ υποσχόμενο αποτέλεσμα ε, που απορρέει από τη χρήση νέων τεχνικών μέσω των οποίων μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Επίση, οι βιολογικοί καλλιεργητέ που επισκέφθηκαν τα δικά μα χωράφια ε, τα τελευταία έξι χρόνια ε, έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό. Φυσικά υπάρχουν διάφορα είδη βιολογικών καλλιεργητών, αλλά πώς να το πω, οι πιο προοδευτικοί μεταξύ τους, για να το πω έτσι, ε, βλέπουν πολύ θετικά τη χρήση τεχνικών, ίσως όχι αυτή συγκεκριμένης, αλλά μιας τεχνικής μέσω της οποίας ε, μπορούμε να φτιάξουμε τις καλύτερες δυνατές ποικιλίε ε, που απαιτούν λιγότερο ψεκασμό από ότι απαιτούν αυτή τη στιγμή οι σημερινές καλλιέργειες. Ε, αναμφίβολα επισήμανση, ναι, είναι κάτι απαραίτητο. Όλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ξέρουν τι αγοράζουν και να ξέρουν τι απορρίπτουν. Αλλά ταυτόχρονα φυσικά είναι σαφές ότι εμείς ως ε, κοινότητα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιούμε λιγότερα βιοκτώνα σε όλες τις καλλιέργειες. Και αυτές οι τεχνικές μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή η μόνη λύση αλλά είναι μέρος ίσως της λύσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ, πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Να απαντήσω ορισμένες που σχετίζονται με την επισήμανση και με τη βιοπικιλότητα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών είναι κάτι υποχρεωτικό σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή όμως δεν έχει να κάνει τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια. Μόνο ε, τα γενετικά μεταλλαγμένα φυτά και γενετικώς μεταλλαγμένοι οργανισμοί που έχουν αξιολογηθεί ως ασφαλείς σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και τις σημερινές προόδους ε, βάσει εκτίμησης κινδύνου μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά ως ασφαλή προϊόντα. Η υποχρεωτική λοιπόν επισήμανση είναι απλά ενημερωτική για τους καταναλωτές το ποια ήταν η μέθοδος ε, παραγωγής, ε, το ποια ήταν η πηγή ε, των προϊόντων αυτών είναι άλλο θέμα αυτών των τροφίμων και ζωοτροφών. Επίσης γίνονται πολλές συζητήσεις όχι μόνο στην Ευρώπη περί υποχρεωτικής ή προαιρετικής επισήμανσης κατά την άποψή μου η επισήμανση γίνεται για να έχουν ελεύθερη επιλογή οι καταναλωτές. Ε, οι καταναλωτές πρέπει να καταλαμβάνουν ε, ε, τι σκοπό εξυπηρετεί η επισήμανση και να καταλαβαίνουν και πώς έχουν παραχθεί αυτά τα προϊόντα. Να σας πω και δύο ενημερωτικά πράγματα για τη βιοπικιλότητα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, τα γενετικώς μεταλλαγμένα ε, και οι άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούμε όπως οι δείκτες, ε, η υποβοηθούμενη επιλογή, το genotyping, οι συμβατικές τεχνικές όλα αυτά είναι απλά εργαλεία. Δεν υπάρχει πανάκια. Δεν υπάρχει μία ενιαία τεχνική η οποία λύνει όλα τα προβλήματά μας. Και επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι θα εμφανιστούν και νέες τεχνικές στο μέλλον. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση της αντίστροφης βελτίωσης. Ε, η αντίστροφη βελτίωση δεν είναι απλά μια τεχνική, είναι μια έννοια, μια ιδέα επιστροφής στα γονίδια που έχουν χαθεί μέσα στα χιλιάδες χρόνια ε, επιλογής, ε, φαινοτυπικής επιλογής να βρούμε δηλαδή τα γονίδια που χάθηκαν μέσα στην εξέλιξη και να τα ενσωματώσουμε όχι διασταυρώνοντας τα μέσα στις νέες μόνο αλλά χρησιμοποιώντας και μοριακές μεθόδους. Χάρη λοιπόν στις μοριακές τεχνικές σήμερα μπορούμε να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα των φυτών ή άλλων οργανισμών και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωσή τους. Όταν μιλάμε για βιοπικιλότητα επίσης, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βιοπικιλότητα στις περισσότερες περιπτώσεις σχετίζεται με τα διαφορετικά περιβάλλοντα. Δεν έχουμε βιοπικιλότητα στα δικά μας χωράφια. Ε, αν υπάρχει εκεί τότε έχουμε γενετική βιοποικιλότητα. Αν καλλιεργούμε την ίδια ποικιλία με το ίδιο γενετικό υπόβαθρο σε μεγάλη κλίμακα, αυτό δεν αποτελεί ε, γενετική ε, ποικιλία. Το θέμα λοιπόν δεν είναι πόσα πολλά διαφορετικά είδη έχουμε, αλλά και που τα βρίσκουμε. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα είναι να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα επιτόπου μέσω της ε, εντατικοποίησης της ε, παραγωγής ορισμένων καλλιεργειών σε ορισμένες περιοχές και αφήνοντας τα φυσικά συστήματα, τα συστήματα της φύσης να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Οπότε, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις... Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην εκπρόσωπο από την Γενική Διεύθυνση Υγείας. Αν φυσικά επιθυμεί το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Όπως είπατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με μια ερμηνεία των εφισταμένων κειμένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρη συνείδηση και επίγνωση του τεράστιου δυναμικού των νέων τεχνολογιών, του δυναμικού για την έρευνα, για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου και της ευρωπαϊκής γεωργίας. Βέβαια, υπάρχει ένα κείμενο η οδηγία 2001 κάθετος 18 που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η οδηγία αυτή περιέχει ορισμό των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, αναφέρει τις τεχνικές που οδηγούν σε γενετική μετάλλαξη, τεχνικές που δεν οδηγούν σε γενετική μετάλλαξη, σε τεχνικές που ναι μεν οδηγούν σε, σε γενετική μετάλλαξη, αλλά παρόλα αυτά εκπίπτουν του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας. Αυτή την ε, οδηγία την εξετάζουμε, προβαίνουμε σε μία νομική ανάλυση, ώστε να δούμε αν οι νέες τεχνικές, η Genesis, ε, οι τεχνικές διόρθωσης του γονιδιώματος, οι άλλες τεχνικές, οι νέες τεχνικές αυτές, ε, εξετάζουμε και προσπαθούμε να εξακριβώσουμε κατά πόσο εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη ισχύουσα νομοθεσία. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται νομική ανάλυση εδώ. Και αυτό το χαρακτήρα θα έχει η συγκεκριμένη ανάλυση, τον νομικό. Αν μία τεχνική οδηγήσει στη, σε μία γενετική μετάλλαξη που δεν εξαιρείται από την οδηγία, σημαίνει ότι χρειάζεται επισήμαση και έλεγχος. Φυσικά δεν είναι άμερη συνεπειών μια τέτοια λύση, ένας τέτοιος χαρακτηρισμός. Γιατί έχουμε πολύ αυστηρές διατάξεις για τις γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι βέβαια τους κρίνουν πολύ χαλαρούς. Εμείς θεωρούμε ότι είναι αυστηρό το σύστημα για τα γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα και ε, είναι πολύ δαπανηρή η υποχρέωση που ε, επιβάλλεται από την νομοθεσία για κάποιον που θέλει να θέσει σε εμπορία τέτοια προϊόντα. Και μόνο οι μεγάλες πολυεθνικές μπορούν να λάβουν τέτοιο κόστος. Οπότε αν μερικές τεχνικές πέσουν στο πεδίο εφαρμογής των γενετικών τροποποιημένων, οργανισμών θα είναι τεράστιο το κόστος γιατί θα χρειαστεί επισήμαση. Θα πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα ότι πρόκειται για γενετικό μεταλλαγμένο οργανισμό και αυτό δεν είναι σίγουρα καλό για την προβολή του, δεν θα σπεύσει ο κόσμος να το αγοράσει, γιατί στην Ευρώπη στα τρόφιμα προορίζονται σε ανθρώπινη κατανάλωση, ο χαρακτηρισμός ε, του μεταλλαγμένου τροφίμου δεν βοηθάει την πρόθεση του προϊόντος. Βέβαια, όταν ε, τα γενετικώς τροποποιημένα αφορούν τις ζωοτροφές, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη νομική αξιολόγηση των ε, νέων τεχνικών. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα την ολοκληρώσουμε μέχρι τα τέλη του έτους. Δύσκολο το βλέπω. Παρ' όλα αυτά, ο Επίτροπος είπε τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας ότι εντείνουμε τις προσπάθειές μας και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να σας υποβάλουμε κάποια πορίσματα σε αρχές του επόμενου έτους τουλάχιστον, ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Μάλιστα, πρόκειται να συγκροτήσουμε και μία ομάδα εμπειρογνωμόνων με παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών και μάλιστα οι ευρωβουλευτές μαζί ζήτησαν συμμετοχή σε αυτή την ομάδα. Θα προσκαλέσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν, πάντως θα προσκαλέσουμε σε αυτή την ομάδα των εμπειρογνωμόνων και θα έχουμε διαβούλευση και με τους ε, διαφόρους συντελεστές, τους ενδιαφερομένους. Αφού ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η νομική αξιολόγηση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δούμε τι συνέπειες θα προκύψουν. Ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν με το πόρισμα αυτό και θα εφαρμόσουν τις συστάσεις που θα προκύψουν από την νομική ερμηνεία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποια στιγμή σε αρχές του επόμενου έτους θα αποκατασταθεί αυτή η ασφάλεια του δικαίου, γιατί όλοι είπαν ότι πρόβλημα για τον κόσμο και για την βιομηχανία είναι αυτό το νεφέλωμα, όταν δεν ξέρει κανείς τι να περιμένει. Χρειάζεται διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου. Φυσικά ασφάλεια δικαίου δεν θα ικανοποιήσει τους πάντες. Μερικοί θα δυσαρεστηθούν, αλλά σίγουρα θα πρέπει αυτή η νομική αξιολόγηση να ολοκληρωθεί με σοβαρό τρόπο και στις αρχές του επόμενου έτους κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το πρώτο τμήμα της δημόσιας μας ακρόασης. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τους δύο πρώτους καλεσμένους μας. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης και καλώ τους ε, τρεις επόμενους εμπειρογνώμονες να λάβουν θέση. Θα έχουμε τώρα την ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερομένους για τα πολύ αυτά σημαντικά θέματα που είναι το αντικείμενο της σημερινής δημόσιας ακρόασης. Πρώτος ομιλητής στο δεύτερο τμήμα θα είναι ο κύριος Γκάρλιχ Φον Έσεν, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Παραγών Σπόρων, ΕΣΑ. Θα μιλήσει για 10 λεπτά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση Σπόρων είναι η φωνή της Ευρωπαϊκής ε, Βιομηχανίας Παραγωγής Σπόρων. Ε, συμμετέχουν σε, αυτό, σε αυτήν 35 εθνικές ε, οργανώσεις και από τα κράτη-μέλη αλλά και από τρίτες χώρες και εκπροσωπεί χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου καθώς και 70 εταιρείες ή ε, άμεσα ασχολούμενες με την παραγωγή ή συναφείς με τον κλάδο των σπόρων. Έχετε το λόγο κύριε Φων Έσεν. Thank you, Chairman, and, uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής σας εγγράψατε το σημαντικό αυτό θέμα στην ημερησία διάταξή σας και μας δίνει την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε. Ήδη έχετε στην εισαγωγή σας πει ορισμένα πράγματα. Ο τομέας σπόρων στην Ευρώπη είναι αρκετά ποικίλο, έχει επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, πολλές μικρές και μεσαίες και πολλές μικρές επιχειρήσεις, είτε Αυτές αναμειγνύονται σε παραγωγή σπόρων και σε βελτίωση φυτών ή ορισμένες κάνουν μόνο τη διάθεση στην αγορά, το marketing. Κάθε χρόνο δημιουργεί ο κλάδος 3.500 νέα προϊόντα, νέες ποικιλίε που είναι διαθέσιμες βεβαίως από όλα τα είδη στους ε, αγρότες. Και μέχρι τώρα έχει σημειώσει 40.000 νέα είδη, ή ποικιλίες μάλλον, ε, στη, στο κατάλογο, στους καταλόγους του. Μεγάλη επιλογή και μεγάλη προσφορά. Ρωτούν πολλοί αν μπορούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αγροπικιλία. Αλλά βέβαια αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει δηλαδή επιλογή. Τα γεγονότα τώρα. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Γνωρίζετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Χρειάζεται να μπορούμε να παράγουμε περισσότερα, πολύ περισσότερες ε, ποσότητες τροφίμων για να μπορέσουμε να ταΐσουμε ολόκληρο τον κόσμο. 80% της βελτίωσης της αποδοτικότητας της γεωργίας οφείλεται σε βελτιωμένα genetics. Βλέπετε και το πίνακα, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Είναι πάντως λογικό να πει κανείς ότι προσπαθούμε να μειώσουμε όσο γίνεται την χρήση ε, ζυζανιοκτώνων και άλλων παραγόντων παρά τις αλλαγές του κλίματος και παρά άλλους περιοριστικούς παράγοντες έχουμε μπορέσει ωστόσο να αυξάνουμε την αποδοτικότητα της παραγωγής genes and brains που έχουμε εδώ διαθέσιμα στην Ευρώπη. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι οι βελτιώσεις φυτών χρειάζεται πολύ χρόνο. Κατά μέσον όρο, όπως είπαν και οι δύο καθηγητές πριν, 10 έως 15 χρόνια μέχρι του φτάσει μια νέα ποικιλία στην αγορά. Αυτό δεν θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στο μέλλον. Χρειάζεται να βελτιώσουμε την προσπάθεια αυτή αλλά και να την επιταχύνουμε πολύ. Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι που προωθεί ο κλάδος σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς προσπαθούμε να το κάνουμε ένα σημαντικό πράγμα είναι να πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον μονάχα ευρωπαϊκή ή αμερικανική νότια νότιο-αμερικανική σπόρη. Οι σπόροι διακινούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, διαρκώς. Επίσης, ε, οι ε, γονιδιαματικές ποικιλίε μετακινούνται παντού σε όλο τον κόσμο. Ορισμένα που βρίσκουμε εδώ στην Ευρώπη τώρα έρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα ευρωπαϊκό καλάθι ή ένα, ευρωπαϊκό, ή ένα αμερικανικό και ούτω καθεξής. Δεν είναι πλέον ερμητικά κλειστά τα πράγματα αυτά. Επομένως, οι σπόροι μετακινούνται παντού για να επιταχύνουν τις διαδικασίες παραγωγής. Όμως, αυτό δεν φτάνει. Αυτό που βλέπετε επίσης είναι ότι αναπτύσσουμε και νέα γνώση γινόμαστε ευφιέστεροι, γνωρίζουμε περισσότερα για το πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία βελτίωση των φυτών, ποια εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πώς αντιδρούν τα φυτά και όλα αυτά μας έχουν επιτρέψει να επιτύχουμε σημαντικές πρόοδους και ορισμένα από τα βήματα των πρόοδων αυτό τα βλέπετε στη διαφάνεια. Έχουμε λοιπόν και άλλα εργαλεία στην εργαλειοθήκη μας. Γινόμαστε λοιπόν σοφότεροι, γνωρίζουμε καλύτερα τι μπορούμε να επιτύχουμε και πώς. Γινόμαστε ακριβέστεροι και πιο αποφασισμένοι να επιτύχουμε τις ε, ακριβείς αλλαγές στο γονιδιώμα. Η βασική λοιπόν ερώτηση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα και την αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτές οι τεχνικές είναι GM, είναι δηλαδή ε, ε, γενετικό, γενετική τροποποίηση ή όχι. Είναι σημαντικό το ερώτημα αυτό. Η πρώτη απάντηση που δόθηκε είναι ότι όντως η ερώτηση αυτή είναι σημαντική. Οι τεχνικές αυτές είναι που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ή όχι. Σύμφωνα με το JSRC, όλες αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, από όλων των ειδών της επιχειρήσης. Δεν μιλούμε εδώ για business technology. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα και από μικρούς ε, αγρότες και από, από μικρούς ε, ε, επιχειρηματίες και για μικρές παραγωγές σχετικά έχει σημασία κοινωνικο-οικονομική. Βεβαίως, ναι, έχουν τεχνικές αυτές πολύ μεγάλη κοινωνικο-οικονομική σημασία για τον τομέα της βελτίωσης των φυτών και βεβαίως και σε ολόκληρη την αλυσίδα. Ιδίω βέβαια για τους πελάτες μας, τους αγρότες δηλαδή που παράγουν φυτικές εσοδίες, αλλά και μέχρι το τελικό καταναλωτή. Υπάρχει και πολύ τεχνολογικό δυναμικό, διότι επιτρέπει οι τεχνικές αυτές να είναι ακριβείς και να ευθυγραμμίζεται το ότι μπορούμε να κάνουμε τεχνικά με αυτά που επιθυμούν να δουν οι καταναλωτές. Αυτό που κάνουμε δηλαδή είναι να γινόμαστε υπό την πίεση των καταναλωτών ακριβέστεροι και ταχύτεροι. Και αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο σημείο. Πού βρισκόμαστε τώρα οι νομικές ερμηνείες. Δηλαδή αυτές οι τεχνικές εμπίπτουν μέσα στον ορισμό των ε, γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών ή τροποποιημένων οργανισμών. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα έχει εξετάσει αυτά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει καταλήξει το συμπέρασμα μετά από τέσσερα χρόνια δουλειά ότι η πλειονότητα των τεχνικών αυτών δεν απαιτούν κανόνες του είδους των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ορισμένες ωστόσο ναι, απαιτούν σύμφωνα πάντως με τις απόψεις αυτών των εμπειρογνωμών των των χωρών μελών. Αυτά σύμφωνα με μια μελέτη του 2012. Από τότε και έχουν γίνει και άλλες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα και οι πιο πρόσφατες αναφέρθηκαν πριν. Και βεβαίως και από τις γερμανικές αρμόδιες αρχές έχει έχουν επιβεβαιωθεί τα αποτελέσματά τους. Ένα σημαντικό θέμα είναι και η δυνατότητα επιβολή. Δηλαδή θα πρέπει να νομοθετεί κανεί πράγματα τα οποία μπορεί και να επιβάλλει. Πάλι εμπειρογνώμονες των χωρών μελών λένε ότι δεν μπορούν τελικά να διακρίνουν το αποτέλεσμα των τεχνικών αυτών, το προϊόν, το τελικό προϊόν δηλαδή, από αυτό που προκύπτει από την φύση. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, δεν θα μπορούμε να απαγορεύσουμε, απαγορεύσουμε και δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο εάν τελικώς παράγουμε τα ίδια προϊόντα όπως η φύση με λίγη τεχνική βοήθεια. Πού βρισκόμαστε λοιπόν τώρα. Εδώ βρισκόμαστε. Ελπίζω ότι είμαστε πια κοντά στο να εξαλείψουμε αυτές τις ασάφειες βάζοντας σταυρουλάκια σε ορισμένα τετραγωνάκια έτσι ώστε τελικά να επιτρέψουμε να είναι προσβάσιμες οι τεχνικές αυτές και τα προϊόντα αυτά σε όλους τους γεωργούς για προς όφελος και της κοινωνίας και της γεωργίας και της ασφάλειας παραγωγής τροφίμων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Επόμενος καλεσμένος μας είναι ο κύριος ε, Χέκερ, ο πρόεδρος της πλατφόρμας για τις νέες τεχνικές βελτίωσεις. Θα μας μιλήσει για τα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι μόνο. Ε, η πλατφόρμα του είναι μια, ένα συνασπισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων και ε, κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητικών Ινστιτούτων που μεταξύ άλλων προσπαθούν να αποσαφηνίσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο των νέων τεχνικών βελτίωσης. Και μάλιστα ο κ. Χέκερ έχει πλούσια εμπειρία στη Γεωργία και κυρίως ε, στο Ολλανδικό Υπουργείο Γεωργίας. Κύριε Χέκερ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε και κύριοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος. Ευχαριστώ, επαναλαμβάνει ο μιλητής κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, ε, μέλη του Κοινοβουλίου. Μπορεί να επαναλάβω κάποια πράγματα που υπόθηκαν ήδη, αφού είμαι ο τέταρτος βέβαια. Οπότε θα περάσω τις ε, διαφάνειες ε, σχετικά γρήγορα. Οι νέες τεχνολογίες, ε, η πλατφόρμα NBT έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το ζήτημα των νέων τεχνολογιών βελτίωσης. Για ποιο λόγο, διότι ο τομέας βελτίωσης των φυτών βασίζεται σε καινοτόμες λύσεις για να παραμείνει ανταγωνιστικός, όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παγκοσμίω. Λόγω των αυστηρών κανονισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές επιχειρήσεις και πολλές μικρές ε, εταιρείες ε, επένδυσαν ε, πάρα πολύ στην έρευνα και την ανάπτυξη των για τις NBT. Ξέρετε, περίπου το 50% της έρευνας έγινε εδώ στην Ευρώπη για τα NBT, όχι εκτός. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να, διασαφιστεί το, να διασαφανιστεί το κανονιστικό καθεστώς για, αυτά, για αυτές τις NBT διότι η έλλειψη διαφάνειας μπλοκάρει την καινοτομία. Όταν αυτές οι τεχνικές βελτίωσεις ε, ενταχθούν, ε, ε, περιορίζονται από τους κανονισμούς, αποτελούν φόρτο για τον τομέα, σημαίνουν και απώλεια εσόδων και ε, μη δυνατότητα αντιμετώπισης των κοινωνικών ε, προκλήσεων. Εμείς αγωνιζόμαστε για νομική ε, βεβαιότητα, αλλά, παρέχουμε και αλλά και το να παρέχουμε σε όλους επιστημονικές σαφείς πληροφορίες, διότι η πλατφόρμα NBT δεν αφορά μόνο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα βελτίωση των φυτών, περιλαμβάνει και μέλη μεταξύ γνωστών ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Ο τίτλος της ε, παρουσίασης μου όμως είναι «Κοινωνικές ε, προκλήσεις». Εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνικές είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Μέχρι το 2050 θα φτάσουμε πληθυσμό 9 δισεκατομμυρίων και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τραφούν κάπως. Οι πόροι που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν. Ε, περίπου το 70% όλου του νερού ε, χρησιμοποιείται από ανθρώπους ε, στον, τομέα, στον αγροδιατροφικό τομέα και λόγω των κλιματικών αλλαγών απειλείται η διατροφική ασφάλεια. Οπότε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις επιστήμες. Το θέμα δεν είναι αν θα χρησιμοποιήσουμε τη γενετική, αλλά ποια γενετική για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κοινωνικά προβλήματα. Ας είμαστε σαφείς. Ε, η βελτίωση των φυτών ξεκίνησε πριν από 9-11 χιλιατηρίδες. Δεν είναι κάτι νέο. Απλά συνεχίζουμε τις τεχνολογίες ε, επιλέγοντας ε, τα φυτά ουσιαστικά, ουσιαστικά με, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Για να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές, τα κοινωνικά προβλήματα χρειάζεται να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των πόρων, χρειαζόμαστε υψηλότερη αντίσταση σε επιβαρυντικούς παράγοντες για όλων των ειδών τα φυτά, ε, γρηγορότερες διαδικασίες βελτίωσης ε, και πιο αποτελεσματική βελτίωση. Με αυτές τις νέες ε, τεχνολογίες βελτίωσης μπορεί να αυξήσουμε την παραγωγή μειώνοντας έτσι τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης κάνουμε πιο αξιόπιστες τις καλλιέργειες για τους γεωργούς και συμμορφωνόμαστε με ε, πρότυπα υψηλότερη ε, ποιότητα ε, διατροφική όσον αφορά τα διατροφικά απόβλητα και, και οπότε καλύτερο για του καταναλωτέ και για τη φύση. Οπότε οι NBT μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν πολλά κοινωνικά προβλήματα, αλλά το νομικό πλαίσιο είναι ασαφέ και εμεί το παλεύουμε εδώ και 8 χρόνια. Όλα ξεκίνησαν με την οδηγία 2018 και πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η οδηγία βασίστηκε σε συγκεκριμένες διαδικασίες, αλλά εμείς την μελετήσαμε. Αλλά ξέρετε, δεν βασίζεται μόνο σε διαδικασίες, βασίζεται και σε προϊόντα ουσιαστικά. Αν πάρει κανείς τον ορισμό, εδώ βλέπουμε 7 ε, ερωτήσεις. Είναι οργανισμός, δεν είναι άνθρωπος, ε, έχει αλλοιωμένο γενετικό υλικό, η γενετική αλλοιώση δεν συμβαίνει φυσιολογικά, η γενετική τροποποίηση συμβαίνει τουλάχιστον μέσω της χρήσης των τεχνικών που παρατίθεται στο παράρτημα 1α μέρος 1, η τεχνική δεν παρατίθεται στο παράρτημα 1α μέρος 2 και η τεχνική δεν παρατίθεται στο παράρτημα 1β. Πρέπει κανείς να απαντήσει όλες αυτές τις ερωτήσεις καταφατικά, αλλιώς το προϊόν δεν είναι γενετικώς μεταλλαγμένο. Τι κάναμε λοιπόν στην πλατφόρμα. Φτιάξαμε ένα διάγραμμα ροής βάσει αυτών των 7 ερωτήσεων. Οι τέσσερις ερωτήσεις ε, βασίζονται στο προϊόν και οι άλλες τρεις στις διαδικασίες. Φυσικά είναι πολύ μικρά η γραμματοσυρά εδώ για να τη διαβάσετε, αλλά πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας μας όπου μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το έγγραφο όπου για κάθε ναι, τεχνική, κάναμε ένα τέτοιο διαγράμμα ροής και εκεί μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του γιατί ορισμένες από αυτές τις τεχνικές δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας για τα ε, μεταλλαγμένα ε, και άλλες, ναι. Ξέρετε, ο τομέα είναι καινοτόμο. Έχει κύκλο εργασιών 45 δι το 2012. Δημιουργεί πολλέ θέσει εργασία ε, εξειδικευμένε, συχνά εκτό των αστικών περιοχών. Οπότε πολύ σημαντικό για πολλέ περιοχέ τη Ευρώπη. Είναι επίσης ένας τομέας ε, με πολύ ψηλές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Σχεδόν το 15% έως το 25% του κύκλου εργασιών επενδύεται στην έρευνα και την ανάπτυξη. Τι κάναμε λοιπόν με το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, κάναμε μια μελώδη για να δείξουμε τις τα κοινωνικά αποτελέσματα και χρησιμοποιήσαμε όλη την αλυσίδα, όχι μόνο τους βελτιωτές, αλλά και τους γεωργούς, τους παραγωγούς, μέχρι τους καταναλωτές. Όλοι επηρεάζονται από αυτές τις νέες τεχνικές. Ε, και φυσικά για τους βελτιωτές ε, φυτών είναι πολύ σημαντική η ακρίβεια και η ταχύτητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπολογίζουμε τα, από τις επιπτώσεις από την ε, απώλεια έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα βελτίωσης των φυτών. Όπως είπα, ε, η βιομηχανία σπόρων έχει κύκλο εργασιών 8,5 δις με επίπεδο 10% στην έρευνα και την ανάπτυξη και η συνολική επενδυτική αξία είναι σχεδόν 860 εκατομμύρια ετησίως. Απόλυα 30% στην έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει απώλεια επένδυση σε εξοπλισμό υψηλού επίπεδου και θέσει εργασία αξία περίπου 258 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα και για του ε, αγρότε. Και αυτοί χρειάζονται υψηλότερη αντίσταση σε βιωτικού και αβιωτικού παράγοντε επιβάρυνση, βελτίωση τη αποτελεσματικότητα γεών και πόρων, βελτίωση ε, τη αποτελεσματικότητα ε, τη συγκομιδή και μείωση του φορτίου σύνδεση. Το δεύτερο παράδειγμα σχετίζεται με την αντίσταση στον περονόσπορο. Ήδη έχουν δοθεί, δόθηκε από τον προηγούμενο ομιλητή η σχετική ενημέρωση. Όταν ψεκάζει κανεί μόνο δύο-τρει φορέ το χρόνο αντί για δέκα, εξοικονομεί πολλά χρήματα. Εμεί υπολογίσαμε ότι οι αγρότε έτσι θα εξοικονομούσαν σχεδόν 900 εκατομμύρια ευρώ μόνο εντό Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την ε, έλλειψη ανάγκη ε, ψεκάσματο. Και φυσικά αυτό έχει τεράστια ωφέλη και για τους καταναλωτές και για το περιβάλλον. Μετά όσον αφορά τους παραγωγούς τροφίμων και τους λιανοπολιτές, οι παραγωγοί μπορούν να βελτιώσουν τις απαιτήσει ε, παραγωγής, έτσι διευκολύνεται η ζωή τους με λιγότερα απόβλητα κατά τη διαδικασία παραγωγής. Αλλά επίσης έχουμε και μεγαλύτερη ποικιλία των προϊόντων, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, διάρκεια αποθήκευσης και λιγότερα συνεπώς τροφικά απόβλητα. Είμαι πολύ γρήγορος. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τον υπολογισμό για τη μείωση των ε, διατροφικών αποβλήτων, η Επιτροπή εκτιμά ότι στην Ευρώπη πετάμε περίπου 90 εκατομμύρια τόνου τροφίμων ετησίων, που μπορεί να φτάσουν του 120 εκατομμύρια τόνου το 2020. Αυτό θα σήμαινε ότι αν είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευση μέσω αυτών των νέων τεχνικών, θα μπορούσαμε να έχουμε 10% απόβλητα, δηλαδή μείωση 9 εκατομμυρίων τόνων. Δηλαδή αυτό αντιστοιχεί σε 40 σχεδόν δισεκατομμύρια ε, ευρώ, 36 ε, ε, ετησίως και, και λιγότερες εκπομπές κατά 36 εκατομμύρια τόνους. Είναι καταπληκτικό λοιπόν αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε με αυτές τις νέες τεχνικές. Και ο καταναλωτής επίσης θέλει το φαγητό του να είναι πιο υγιεινό, να έχει καλύτερες βιταμίνες, λιγότερα αλλεργιογόνα κτλ. Αλλά θέλει και καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στα τρόφιμα, το χρώμα, την οσμή, όλα αυτά μπορούν να ενισχυθούν με αυτές τις τεχνικέ. Φτάνοντας στο τέλος παρουσιασή μου, θέλω να πω δύο πράγματα. η υπερβολική, ο κανονικός, κανονιστικός υπερθεματισμός και οι καθυστερήσει στη χάραξη πολιτικής ε, θα οδηγήσουν στο εξωτερικό τους βελτιωτές των φυτών για να βρουν άλλες ερευνητικέ εγκαταστάσεις και επενδύσεις. Έχουμε ήδη παραδείγματα. Τέτοια μικρές εταιρείε ε, θα αντιμετωπίσουν σοβαρή μείωση της αξίας τους με τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν τελείως τις δραστηριότητες τους ε, όταν δεν έχουν αρκετά χρήματα για να αντεπεξέλθουν στα κανονιστικά συστήματα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα σήμαινε και απόλυτη ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τι εταιρείε που βρίσκονται εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, όταν οι κανονισμοί είναι πιο απλοί και το κανονιστικό πλαίσιο είναι πιο σαφές, οι επενδύσεις στην ε, έρευνα και την ανάπτυξη θα παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επηρεάσουν θετικά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Όχι μόνο στον τομέα της βελτίωσης των φυτών, αλλά σε ολόκληρη την αλυσίδα. Τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και όπως αναφέραμε ήδη η ανείχνευση τέτοιων προϊόντων είναι κάτι πολύ δύσκολο δηλαδή και για το εμπόριο θα ήταν μεγάλο το πρόβλημα αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι με μείωση των κανονιστικών περιορισμών θα βοηθήσουν οι τεχνικές αυτές την αντιμετώπιση πολλών κοινωνικών προβλημάτων για ένα πιο αιφόρο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε. Και τώρα περνάμε στον τρίτο μας εμπειρογνώμονα, τον κύριο Κρίστοφ Τεν, που είναι εκτελεστικός διευθυντής του Test Biotech. Θα μας μιλήσει 10 λεπτά για τεχνικά και νομικά επιχειρήματα που αφορούν την διόρθωση του γονιδιώματος και τη βελτίωση των φυτών. Ε, ο κύριος Στέν είναι εκτινίατρος και για 20 χρόνια ασχολείται με θέματα βιοτεχνολογίας. Η Test Biotech είναι μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιεί μελέτες επιπτώσεων σε θέματα βιοτεχνολογίας, έρευνα, ε, ανάλυση ε, δεοντολογική, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων και αξιολόγηση κινδύνων στην υγεία και στο περιβάλλον. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Θα περάσω κατευθείαν στην παρουσίασή μου. Όπως είπατε, προσπαθούμε να κρατήσουμε την ανεξαρτησία μας από, την, από τον κλάδο της βιοτεχνολογίας και να στηρίξουμε τα επιχειρήματά μας σε επιστημονικά απορίσματα και αν σας ενδιαφέρει η παρουσίαση έχω φέρει και αντίγραφα, αλλά θα τη δημοσιεύσουμε και στην ιστοσελίδα μας. Σας παραπέμπω εκεί. Τώρα, ποιες είναι οι πιο σημαντικές τεχνολογίες. Είναι θέματα διόρθωσης του γονιδιώματος, με τεράστιο δυναμικό. Πρόκειται για την αλλαγή του γονιδιώματος στο κύτταρο με ε, σύντομο συνθετικό DNA. Αυτή είναι μια τεχνολογία, τα ολιγονουκλεοτίδικα νουκλεοτίδια. Άλλη τεχνική είναι η χρήση νουκλεασών που μπορούν να εκτοπίσουν ή να προσθέσουν γονίδια. Knockout ή knock-in μπορεί κανείς ε, ή να εκτοπίσει γονίδια από συγκεκριμένη θέση ή να προσθέσει. Και επίσης ε, μπορεί κανείς να αλλάξει όχι μόνο τη δομή του DNA, αλλά και τη ρύθμιση του γονιδιώματος. Αυτέ αυτές είναι οι βασικές τεχνολογίες, οι κύριες τεχνολογίες. Δεν χρειάζεται πια να γίνει απομόνωση του DNA από τη φύση. Μπορούμε να έχουμε μια σύνθεση και στο εργαστήριο και να κάνουμε και σχεδιασμό του DNA ακόμη και στον υπολογιστή. Και το δεύτερο που αναφέρονται είναι οι, οι νουκλεάσες ε, για τη διόρθωση του γονιδιώματος. Ε, βρίσκουμε σε συγκεκριμένο σημείο ε, μία δομή. Εκεί μπορούμε να κόψουμε το DNA και είτε να διαγράψουμε είτε να προσθέσουμε γονιδιακή πληροφορία είτε να αφήσουμε το κύτταρο να επιδιορθώσει μόνο του το DNA και που κάναμε τη διακοπή του έλικα. Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές γίνονται συζητήσεις για την νομική ρύθμιση, την κανονιστική ρύθμιση του θέματος αυτού. Ε, είναι εύκολο με την οδηγία του 2018. Υπάρχουν κάποιες παλιές τεχνολογίες που εφαρμοζόταν και πριν τη θέση ισχύ της οδηγίας και έχουμε και νέες τεχνολογίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να τροποποιήσουν τις γενετικές καταστάσεις των φυτών. Αυτές οι τεχνολογίες χρειάζονται ρύθμιση. Πρόκειται για μια προσέγγιση που καθορίζεται από τη διαδικασία και όχι για το, από το κατά πόσο έχουμε νέο DNA ή όχι. Ακόμη και με διακοπή DNA σε συγκεκριμένο σημείο μπορεί να καταλήξουμε σε μεταλλαγμένο οργανισμό. Άρα χρειάζεται ε, ρύθμιση. Οπότε μπορεί είτε να προσθέσουμε είτε να αφαιρέσουμε DNA και αυτό αλλάζει ε, το φυτό και το κάνει διαγωνιδιακό. Βέβαια, μεταλλάξει γίνονται και φυσιολογικά. Πάντω, όταν έχουμε γονίδια από ένα άλλο φυτό, έχουμε διαγωνιδιακό οργανισμό. Το θέμα είναι, υπήρχε τεχνολογία αυτή ενισχύει πριν τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Ε, έχουμε τεχνολογία που επεμβαίνει στο DNA, αλλάζει τη γονιδιακή κατάσταση, τη γονιδιακή ρυθμίση του φυτού. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Και έχουμε εδώ δύο νομικά θέματα, Κρέμερ και Σπρέγκερ, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Το πρώτο ξεκίνησε από μη κυβερνητικέ ε, οργανώσει, το δεύτερο από τι γερμανικέ αρχέ. Τα συμπεράσματα είναι τα ίδια, μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο και είναι σαφή και η νομική ανάλυση που περιλαμβάνουν. Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση, στηρίζεται στη διαδικασία. Και ισχύει φυσικά και η αρχή της προφύλαξης που έχει προτεραιότητα. Πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης. Τώρα, ε, υπάρχει ενδιαφέρον ώστε να αλλάξουμε την προσέγγιση από προσέγγιση που προσανατολίζεται στη διαδικασία σε προσέγγιση που προσανατολίζεται στο προϊόν. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε ένα απόσπασμα μιας δημοσίευσης μιας γερμανικής ε, Ομάδα εμπειρογνωμόνων που λέει ότι οι νέες τεχνικές, οι μελλοντικέ τεχνικές μπορούν να αξιολογηθούν ανάλογα με το νέο χαρακτηριστικό και το τελικό προϊόν και όχι από την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί μια νέα ποικιλία φυτού. Σίγουρα η μέχρι στιγμής ε, ε, νομοθεσία δεν υιοθετεί αυτή την προσέγγιση. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρόταση αντιβαίνει σε αυτή την ε, ισχύουσα προσέγγιση. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, έχουμε άλλη νομοθεσία. Εδώ έχουμε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό Nature και εκεί αναφέρονται κάποιες καλλιέργειες ε, των ΗΠΑ που δεν εμπίπτουν στον κανονισμό γιατί έχουν την προσέγγιση που, ε, δεν περιλαμβάνει την αρχή της προφύλαξης, είναι προσανατολισμένη στο προϊόν και υπάρχουν πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα είτε παλιών είτε νέων τεχνολογιών που δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση. Άρα δεν έχουμε ούτε διαφάνεια, ούτε εχνηλασιμότητα και ουσιαστικά δεν εξασφαλίζουμε και επιλογή στον καταναλωτή. Είναι μια συγκεχημένη εικόνα και κανένα δεν ξέρει πού εμπίπτουν αυτέ οι τεχνολογίε. Δεν θα πρέπει να μιμηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αμερικανικό παράδειγμα, αλλά να έχουμε μια πιο σαφή νομοθετική ρύθμιση. Από την άποψη τη επιστήμης θα πρέπει να δούμε τα πιθανά αποτελέσματα. Ε, knockout ή knock-in, δηλαδή ε, διακοπή και αποβολή εκτοπισμό DNA ή προσθήκη DNA. Θα πρέπει να δούμε τι αποτελέσματα έχει αυτή η τεχνική στο DNA ή να δούμε τι αλλαγές έχουμε στη ρύθμιση στη γονιδιακή ή αλλαγές στη σύσταση του φυτού και πώς αντιδρά το φυτό στο περιβάλλον. Όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν σταδιακά και να μην πούμε απλώς ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε ή όχι. Θα πρέπει να τα δούμε περιπτωσιολογικά και ενδελεχώς. Τώρα, γιατί χρειάζεται ρύθμιση. Ένας από τους λόγους είναι ότι αυτό το βήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Ακόμη και στο πρώτο βήμα έχουμε μια μικρή αλλαγή στο DNA. Αν επαναληφθεί πολλές φορές αυτή η αλλαγή, μπορούμε να έχουμε ένα γονιδίωμα με μικρές ή μεγάλες αλλαγές. Οπότε αν αυτό το εξαιρέσουμε από την νομοθεσία δεν ξέρουμε αν κάποιες τεχνικές κατάντι, κάποιες επαναλήψεις ή κάποιες αλλαγές θα οδηγήσουν τελικά σε εκτεταμένες αναδιατάξεις του γονιδιώματος ή ριζικές αλλαγές του γονιδιώματος. Εδώ έχουμε δύο πολύ ωραίες διαφάνειες. Η μία δείχνει τεχνολογία αμερικανική που λέει ότι μία, δύο, τρει εκατό φορές επαναλαμβάνουμε το πρώτο βήμα και με, ουσιαστικά ξαναγράφουμε το, όλο το γονιδίωμα μόνο με μικρές αλλαγές, μικρές μεταλλάξεις, ελάχιστες αλλαγές στο γονιδίωμα με την επανάληψη αυτού του βήματος προκαλούμε ριζικές αλλαγές στο τελικό προϊόν. Οπότε έτσι μπορούμε να ξαναγράψουμε ουσιαστικά το γονιδίωμα του Homo sapiens και να αναχθούμε στον Neanderthal. Και μάλιστα Τσέρτς και Ρέγκης που είναι από τους πιο σημαντικούς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες ε, στον τομέα αυτό λέει ότι η ίδια τεχνική θα λειτουργούσε και για τον Νεάντερνταλ ε, και θα μπορούσαμε έτσι να αναχτούμε σε αυτό το γονιδίο μας. Ό,τι αφορά το κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο, κάναμε κάποια έρευνα και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά διπλώματα ευρυστεχνία στον τομέα αυτό. Προς το παρόν είναι κάπως και εικόνα. Έχουμε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά όχι μόνο. Ε, και εδώ έχουμε δεσπόζουσα θέση των συνήθων υπόπτων της Dow AgroScience, της Bayer και της Monsanto. Αυτές είναι οι πιο ισχυρές ε, εταιρείε, επιχειρήσεις που έχουν πολλά διπλώματα ευρυστεχνίας και έχουν και κάποιους μικρούς εταίρους. Ε, και φυσικά ισχύει η συγκέντρωση της αγοράς εδώ. Πάντως οι όλες εξελίξεις κυρίως θα, θα οδηγηθούν στις... στα διπλώματα ευρυστεχνίας και θα είναι πιο δύσκολο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση χωρίς ένα σύστημα προστασίας. Οι νέες τεχνολογίες θα έχουν υψηλής προστασίας, κυρίως από τα διπλώματα ευρυστεχνίας. Σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό σύστημα, σε τελική ανάλυση δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αν θεσπιστεί η ρύθμιση, περιμένω να ισχύσει, φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων θα κάνει κάποιες συστάσεις για την εκτίμηση αυτών των φυτών και θα χρειαστεί και μελέτη επιπτώσεων του κινδύνου με βάση της, την καθοδήγηση της συστάση της ΕΦΣΑ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρουμε τι θα, αν θα απαιτηθεί αξιολόγηση τελικά των φυτών. Πάντως, ε, αν κοιτάξουμε τη γενική εικόνα, ε, θεωρούμε ότι το νομοθετικό κόστος θα είναι το λιγότερο. Το, το πρόβλημα θα είναι η, προστασία από τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Δεν θα έχουμε πρόσβαση στι νέε τεχνολογίε για τι μικρέ επιχειρήσει, γιατί θα έχουν μονοπολίσει τα διπλώματα ευρεσιτεχνία οι πολυεθνικέ, οι μεγάλε εταιρείε. Οπότε δύσκολο για τις μικρομεσαίες θα είναι να, θα είναι να επιβιώσουν, δεν έχουν κάλυψη από διπλώματα τεχνίας. Οπότε θέλουμε διανομή της τεχνολογίας θα πρέπει να δούμε το θέμα των διπλωμάτων ευρυστεχνίας. Τώρα, από νομική άποψη χρειαζόμαστε καταγραφή, μελέτη επιπτώσεων, επισήμανση, σαφέστατο αυτό, από τις νομικές υποθέσεις που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής. Από επιστημονική άποψη τώρα υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες ακόμη για τις νέες εξελίξεις. Δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Χρειάζεται λοιπόν αξιολόγηση. Θέλουμε περισσότερη εμπειρία δεν μπορούμε να τα μολύσουμε απλώς στην αγορά και να τα αφήσουμε να πάρουν το δρόμο τους. Χρειαζόμαστε ε, ρύθμιση και κατάντη. Και από κοινωνικο-οικονομική άποψη, το πιο σημαντικό περιοριστικό παράγοντας θα είναι όχι το ρυθμιστικό σύστημα, αλλά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Περάμε στο δεύτερο γύρο των ερωταπαντήσεων. Μπορείτε να θέσετε είτε απευθείας ερωτήσεις στους καλεσμένους μας, είτε να κάνετε σχόλια. Κυρία Χόλμπους είναι η πρώτη που ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι σε αυτό που είπε στο τέλος ο Κρίστοφ Τέν, ότι δηλαδή πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά κυρίως τα διπλώματα ευρεστέχνειας. Ερώτηση. Τι σημαίνει αυτό για τους μικρούς παραγωγούς. Εσείς εξηγήσατε πριν ότι τα γονιδιώματα κυκλοφορούν σε ολόκληρο, τον κόσμο. Αν όμως δεν υπάρχει νομοθετική ρυθμίση, αν δεν υπάρχει επισήμανση και όταν εμφανιστεί ένα τέτοιο γονιδίωμα στην παραγωγή ενός μικρού παραγωγού, εγώ βλέπω εδώ να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Αν δηλαδή τα εξαιρέσουμε από την ρύθμιση και δεν φαίνεται πώς θα εντοπίζονται τα γονιδιώματα. Τώρα για την διαδικασία αδειοδοτήσεων. Η 118-2000 οδηγία, 2001-18 μάλλον, εφαρμόζεται σε ορισμένες εφαρμογές που θεωρούνται ως ασφαλείς. Τουλάχιστον αυτό λέει μέσα στο εκτιμώντας 17. Όμως αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για αυτές τις νέες τεχνικές αφού η τεχνολογία αυτή είναι πολύ πρόσφατη και δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, ούτε αν θα είναι ασφαλής. Εάν τώρα πάλι εξαιρέσουμε τις τεχνικές αυτές από τη διαδικασία αδειοδότησης, πάλι δεν έχουμε ούτε αξιολόγηση του κινδύνου, ούτε monitoring, ούτε διαδικασίες αδειοδοτήσεως. Πώς θα γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αν τα βάλει κανείς αυτά όλα κάτω, βλέπω ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί στο να είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη η οποία δίνει τις άδειες, ότι μπορεί να υποβάλει ρωτήσει στις χώρες μέλη, το δε κοινοβούλιο μένει εκτός της διαδικασίας αυτής, σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Και αναφερθήκατε και στις μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Κύριε Φοντέκερ, εσείς μιλήσατε για το πόσα δισεκατομμύρια αξίζει αυτή η αγορά. Όμως δεν είναι μονάχα τα δισεκατομμύρια. Είναι ολόκληρη οικονομική κλάδη, ολόκληρα συστήματα παραγωγής. Οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι έχουν χρηματοδοτήσει, έχουν φτιάξει ολόκληρο ε, σύστημα για την επισήμανση προϊόντων που να δείχνει ότι είναι ελεύθερα από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και όλο αυτό τώρα πηγαίνει στράφη. Αυτά όλα οδηγούν σε μεγάλη έλλειψη ασφάλειας για τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες. Πώς θα γκρεμίσετε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο το έφτιαξαν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι με δικές τους συνεισφορές. Ευχαριστώ. Δεν ζητά κανείς άλλος συνάδελφος το λόγο. Α, συγγνώμη, ο κύριος Χόισλινγκ. Βέβαια, αν δεν θέλει κανένα άλλο, εγώ θέλω. Για τον κύριο Φωνέσεν, ερώτηση. Γιατί μας εξηγήσατε πόσο ένδοξο αναμένει να είναι, αναμένεται να είναι το μέλλον. Είπα και πριν ότι και προ τα ίδια μας λέγανε. Αν τα πράγματα είναι τόσο ωραία και αποτελούν τόσο μεγάλη πρόοδο και είναι μόνο αμοιβαίως εποφελεί. γιατί είστε αντίθετοι με μια ξεκάθαρη επισήμανση. Γιατί να κρύβετε λοιπόν το προϊόν που έχει προέλθει από τεχνική βελτίωση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάποια δυσπιστία. Υπάρχουν δυσπιστίες αν δείτε τα προϊόντα των τέων τεχνολογιών και δείτε και τις εξελίξεις στη Γερμανία, την ελαιοκράμβη που προήλθε από γενετικά τροποποιημένη ε, διαδικασία τέλο πάντων δεν έχει μεγαλύτερη απόδοση άρα πού βρίσκεται η ωφέλεια. Δηλαδή μιλάμε για γενετική τροποποίηση οργανισμών με άλλα μέσα, ας το πω έτσι, αυτό που μας, αυτά που μας εξηγείται εδώ. Όλα αυτά είναι παλιές ιστορίες με νέο μανδύα. Έχω και μια ερώτηση για την Κομισιόν που είπε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα συμπεριληφθεί στην υπόθεση αυτή. Για κάντε το πιο συγκεκριμένο, διότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι έθεσαν ήδη ερωτήσει. Και η Επιτροπή Γεωργίας είπε ότι θέλει να ενταχθεί στη διαδικασία. Δεν είναι μόνο υπόθεση των χωρών μελών και της Κομισιόν, η θέσπιση νέων κανόνων. Η κυρία Χόιμπουχ έχει δίκιο που λέει ότι είναι κρίσιμο για το μέλλον. Είμαστε λοιπόν επισήμως μέσα, είμαστε επισήμως συνομοθέτες ή απλώς ακούτε τη γνώμη μας. Το ζήτημα εδώ είναι κρίσιμο. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλο κανένα να θέλει το λόγο. Οπότε να δώσω το λόγο στην κυρία Τολότη από τη Γενική Διεύθυνση Σάντε. Παρακαλώ. Oui, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ. Θέλω να σχολιάσω διάφορα σημεία που άκουσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μεταξύ. Πρώτα απ' όλα, εάν οι τεχνικές αυτές εντάσσονταν στο πεδίο εφαρμογής ε, της οδηγίας και θεωρούν τον ε, ε, γενετικώς μεταλλαγμένα, η Κομισιόν θα είχε ζητήσει ήδη από την ΕΦΣΑ να επαληθεύσει ότι οι κατητήρες γραμμές που ισχύουν για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς ε, γενικότερα ισχύουν και για αυτές τις νέες τεχνικές. Ε, ε, θα είχαμε λοιπόν ρωτήσει για το δακτύλο ψευδαργύρου, για το transgenesis, για το cisgenesis, αν ίσχυαν οι υπαρξές ε, κατευθυντήρες γραμμές και η ΕΦΣΑ μας είπε ότι οι κατευθυντήρες γραμμές που υπάρχουν είναι επαρκείς, δεν χρειάστηκε δηλαδή να προσθεθεί κάτι, η αξιολόγηση κινδύνων μπορούσε να ακολουθηθεί κανονικά. Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι η Επιτροπή το κατά πόσο θα συμβουλευτεί η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο τα κρατημέλη. Να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μια νομική ερμηνεία της Κομισιόν, ε, ο τρόπος δηλαδή που ερμηνεύει νομικά η Κομισιόν μια ε, οδηγία Δηλαδή η Κομισιόν θα ερμηνεύσει την νομοθεσία. Και η τελική επεξήγηση μπορεί να γίνει από το δικαστήριο. Δηλαδή θα γίνει μια προσπάθεια ερμηνείας ε, από πλευράς Κομισιόν. Μια απόπειρα ερμηνείας. Ξέρετε κάπου πρόκειται για ένα κείμενο της Κομισιόν. Δεν είναι ένα νέο κείμενο που προκύπτει από συναπόφαση. Ε, είναι μια πρόταση της Κομισιόν όπου λέει προτείνω μια νέα νομοθεσία Αλλάζουμε τον ορισμό των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, ξεκινάμε από το μηδέν, ή τα περιλαμβάνουμε όλα ή τα απορρίπτουμε όλα. Αυτό θα ήταν μια πρόταση της Κομισιόν προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για μια νέα νομοθεσία και φυσικά ο συνομοθέτης στο Κοινοβούλιο θα εμπλεκόταν. Αυτό είναι προφανές. Εδώ όμως μιλάμε απλά για μια ερμηνεία ενός νομικού κειμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε παραπάνω ούτε τίποτα λιγότερο από μια απλή ερμηνεία της Κομισιόν υποσχεθήκαμε και η κυρία Ρόιμπουργκ μας είχε καλέσει σε μια συζήτηση και είχε ζητήσει να συμμετάσχει ε, στην παρουσίαση της Κομισιόν την ημέρα όπου θα γινόταν αυτή η ερμηνεία. Εμείς ε, είπαμε τόσο στο email όσο και στο κοινοβούλιο όσο και στους ενδιαφερόμενους Greenpeace, δηλαδή η μικροπαραγωγή οι Ευρωπαϊκέ ενώσει όλοι αυτοί μα υποσχέθηκαν να παρουσιάσουν αυτή την ερμηνεία τη Κομισιόν. Ωστόσο, δεν μιλάμε για ένα κείμενο που εντάσσεται στο πλαίσιο τη συνωμοθεσία, πρέπει να μια απλή ερμηνεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγγνώμη, δηλαδή που πρέπει να σα το πω φυσικά και θα σα ακούσουμε, αλλά εδώ ε, δεν πάβει να είναι παρά μια ερμηνεία τη Κομισιόν που θα ακολουθήσουν ή όχι όλοι. Ελπίζω, ελπίζουμε να θα ακολουθηθεί και σε τελική ανάλυση το δικαστήριο θα είναι εκείνο το οποίο θα αποφασίσει αν η ερμηνεία μα ήταν σωστή ή όχι. Ε, Επίτροπος το ανέφερε, θα ε, ε, εργαστούμε σοβαρά εάν κάποιο προϊόν εντάσσεται στον ορισμό της νομοθεσίας, εντάσσεται. Αλλιώς θα δώσουμε διευκρίνηση. Θα είναι λοιπόν σοβαρή, αυτόνομη η εργασία αυτή, αλλά επαναλαμβάνω δεν πρόκειται παρά για μια ερμηνεία υπάρχοντος κειμένου. Δεν προτείνουμε νέα νομοθεσία μόνοι μας από τη γωνία από τη γωνία μας. Δεν κάνει τέτοια πράγματα η Κομισιόν, ούτε καν έχει εξουσία για τέτοια πράγματα. Άκουσα για την αιτιολογική σκέψη 17. Φυσικά είναι ένα από τα πράγματα που αυτή τη στιγμή αναλύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το έχουμε υπόψη μας, αυτή την αιτιολογική σκέψη. Κατά τα άλλα, Ξέρετε, αλλιώ η, η συζήτηση υπάρχει κίνδυνο να γίνει υπερβολικά τεχνική, οπότε θα σταματήσω εδώ. Ε, λοιπόν, η ομάδα προγνωμόνων θα πρέπει να συνέλθει κατά την άποψή μου, αν όλα πάνε καλά, το Φεβρουάριο. Αλλά δεν ξεχνάμε το αίτημα του Κοινοβουλίου σε καμία περίπτωση να συμμετάσχει στις συζητήσεις αυτές. Δεν το έχουμε ξεχάσει. Θα γίνει, θα συνεδριάσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Οπότε εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν. Α, και η κυρία Σένερα στο μεταξύ βλέπω να ζητάει το λόγο όμως. Después de la intervención de la Comisión... Μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προβληματίζομαι με ανησυχή που επικαλείται το επιχείρημα της νομικής ερμηνείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι αρκετά σοβαρό το θέμα και ουσιαστικό και χρειάζεται εμβριθή συζήτηση. Και περίμενα από τη Βιοτέκ μια διαφορετική άποψη και χαίρομαι που είχαμε και τον καλεσμένο από εκεί. Θα ήθελα να είμαστε πιο πλουραλιστές, γιατί από τους πέντε που μίλησαν οι τέσσερις ακολούθησαν την ίδια άγουσα. Εγώ θα ήθελα να έχουμε μια μεγαλύτερη πολυφωνία στις ακροάσεις μας, για να μπορούμε ε, να έχουμε καλύτερη γνώση και πιο τεκμηριωμένη πριν αποφασίσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους καλεσμένους μας, αν θέλουν, από τρία λεπτά ο καθένας για να απαντήσουν. Οι καλεσμένοι μας παρακαλώ, αν θέλουν το λόγο για να απαντήσουν, έχουν τρία λεπτά ο καθένας. Ποιος θέλει πρώτος το λόγο. Uh, Ο κύριος Στεν... Α, κατάλαβα ότι εγώ πρέπει να λάβω πρώτα το λόγο. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν για την ασφάλεια δικαίου για τους γεωργούς, για την εχνηλασιμότητα και η εφαρμογή της επισήμασης και η εχνηλασιμότητα είναι όλα ανοιχτά θέματα. Πάντως η παραγωγή σπόρων γνωρίζουν ποια προϊόντα καλύπτονται από τι νέε τεχνολογίε και ποια καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνία. Οπότε υπάρχει δυνατότητα λασιμότητα και επισήμανση, αν υπάρχει τέτοια βούληση. Δεν είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Επίση, ε, για την ανάλυση του DNA δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν είχαμε τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτό είναι κάτι που μας το επισήμανε ο κλάδος αλλά δεν στηρίζεται σε επιστημονικά πορίσματα. Πάντως ίσως ήταν δύσκολο σε ορισμένες περιπτώσεις ε, να γίνει ο εντοπισμός μόνο με βάση ανάλυση του DNA. Πάντως κανεί, μπορεί αν θέλει η νομοθεσία να επιβάλλει επισήμανση και χνηλασιμότητα. Τώρα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εκεί χρειάζεται ασφάλεια δικαίου. Γιατί το θέμα είναι ε, αν οι τεχνολογίες διορθώνουν το γονιδίωμα ή είναι τεχνολογίες ε, συμβατή βελτίωσης. Πάντως, ε, ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας μερικές φορές ξεπερνούν το διόρθωση του γονιδιώματος. Καλύπτουν ακόμη και παραδοσιακή βελτίωση. Αναφέρεται ότι όλα τα φυτά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καλύπτονται από το δίπλωμα ευρυστεχνία, άσχετα με το πώ παράγονται. Οπότε είναι σημαντικό εδώ το θέμα. Αν θέλετε να κάνετε διάκριση μεταξύ συμβατική βελτίωση και των νέων τεχνολογιών διόρθωση του γονιδιώματο ε, για, τα διπλώματα ευρυστεχνία, θα πρέπει να το διευκρινίσετε. Γιατί με το ισχύον σύστημα δεν είναι προφανέ ούτε σαφέ. Θα πρέπει να γίνεται διάκριση με το νέο σύστημα μεταξύ παραδοσιακή ε, βελτίωσης και βελτίωσης από διόρθωση του γονιδιώματος και νέες τεχνικές. Δεν ξέρω πόσα λεπτά είπατε. Τρία. Έχω ακόμη ένα. Ε, επίσης, ε, αν δούμε λίγο και το μέλλον, βλέπουμε ότι έχουμε εφαρμογές παρόμοιες με αυτές που γνωρίζαμε. Για παράδειγμα, φυτά ανθεκτικά στα φυτοφάρμακα. Βέβαια, ε, μερικές φορές δεν έχουμε στόχευση των φυτών, αλλά του, του περιβάλλοντος εντόμων, ζυζανίων. Οπότε έχουμε πειρασμό των γονιδιακών συνθηκών όχι μέσα στον αγρό, αλλά και γύρω από τον αγρό. Αυτές οι εφαρμογές πώς θα τις αξιολογήσουμε. Ε, γιατί δεν προσπαθούμε να τις περιορίσουμε μόνο στον αγρό, αλλά οι νέες γενεδιακές πληροφορίες ε, διασπείρονται και εκτός του αγρού και θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να διευκρινιστούν όλα αυτά. Γιατί θέλουμε καλές απαντήσεις για ασφάλεια δικαίου και τη δέουσα προστασία και για τους καταναλωτές και για το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Thank you, Chairman, for uh, the time to... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε λίγο για να απαντήσω. Να απαντήσω σε δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα των αδειών ευρεσιτεχνίας, των διπλωμάτων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Εγώ, ξέρετε, εστιαστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσει. τα μέλη της πλατφόρμας NBT είναι μικρομεσαίες επιχειρήσει, Για αυτές λοιπόν, αυτές οι νέε τεχνολογίες βελτίωσης είναι πολύ σημαντικές. Όπως είπα, σχεδόν το 46% τη έρευνα και της ανάπτυξης γίνεται στην Ευρώπη κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσει ευρωπαϊκές. Για αυτές λοιπόν, για τις ΜΜΕ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειωθεί πρόοδο και να σα δώσω ένα απλό παράδειγμα όταν έχουμε ένα νέο γενετικό τροποποιημένο ε, προϊόν πάει κανείς στο φάκελο στην ΕΦΣΑ και αυτό κοστίζει περίπου 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ. Όταν λοιπόν είσαι μια μικρομεσαία επιχείρηση με κύκλο εργασιών μόνο 20 εκατομμύρια φαντάστε, όπως φαντάστε δεν είναι πολύ δυνατόν να ε, συμμορφωθεί με τον κανονισμό. Οπότε ε, είναι πολύ σημαντικές αυτές τις τεχνικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μουσείο ούτε νησί ε, αυτάρκειας. Ε, ε, είναι κάτι που έχουμε ήδη δει με τα γενικώς μεταλλαγμένα προϊόντα παγκοσμίω. Αυτές οι νέες τεχνολογίες βελτίωσης είναι, ανήκουν στην ίδια περίπτωση. Ορισμένες χώρες ήδη έχουν κάνει κάποια σημαντικά βήματα και έχουν λάβει κάποιες αποφάσεις με αυτές τις τεχνικές για να ε, μην ενταχθούν στον κανονισμό. Οπότε η Ευρώπη πρέπει να δει και τα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία είναι τόσο μεγάλα που χρειαζόμαστε περισσότερα εργαλεία στο προστάσιό μας για να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι τεχνολογίες ε, βελτίωσης ούτε οι τεχνολογίες γενετικής μετάλλαξης. Χρειαζόμαστε και άλλα περισσότερα εργαλεία για να ε, προσφέρουμε καλά προϊόντα μέσω της αγροδιατροφικής ε, ε, αλυσίδα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχουμε τα ίδια προϊόντα σε νέα μπουκάλια. Είναι και τα προϊόντα νέα. Και αν δοκιμάσετε το περιεχόμενο των μπουκαλιών θα δείτε ότι μπορεί να επιλύσει πολλά από τα προβλήματα της κοινωνίας. Yes, thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εγώ να μην μπω σε πολλές λεπτομέρειες της νομικοτεχνικής αυτής της συζητήσεως. Το ερώτημα είναι γιατί φαίνεται να φοβάται τόσο πολύ ο κόσμος αυτή την επιστημονική πρόοδο. Γνωρίζουμε παραπάνω, από, ε, παραπάνω σήμερα για το plant breeding από ό,τι γνωρίζαμε προ πεντακαετίας. Για να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις μεταλλακτικές τεχνικές που θα ε, προσδώσουν στα φυτά τα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε. Γνωρίζουμε πολύ περισσότερα σήμερα. Και φαίνεται να υπάρχει κάποια ομάδα πολιτών, έτσι μου φαίνεται, που θεωρεί ότι η παραπάνω γνώση είναι επικίνδυνη. Όχι, η λιγότερη γνώση είναι επικίνδυνη. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι έχουμε σήμερα. Ε, αποφέρει πολλά πλονεκτήματα η κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί το φυτό και πώς μπορούμε να επιφέρουμε ευεργετικά αποτελέσματα, όχι μόνο αύξηση της παραγωγής, αυτή είναι η κλασική προσπάθεια που θα συνεχίσει να μας απασχολεί, αλλά και ποιοι είναι οι στόχοι. Δηλαδή, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αντοχή, αλλαγή, ε, λιπαρά, βιταμίνες, Δηλαδή μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε παλαιότερα καθόλου ή όπου χρειαζόμασταν πολύ μακρά χρονικά διαστήματα. Και θα μας επιτρέψει επίσης, αν δεν είναι ιδιαίτερα δαπανηρό αυτό, να το κάνουμε και για μικρές παραγωγές, όχι μόνο για το ελαιοκράμβης, όχι μόνο για το καλαμπόκι και όχι μόνο για την πατάτα, αλλά και για πολλά από τα ε, μικρά, μικρές εσοδίες λαχανικών και άλλων. Τέθηκε επίσης η ερώτηση τι γίνεται με την επισήμανση. Δεν θέλετε να το περιλαμβάνετε στην επισήμανση. Ναι, εγώ νομίζω ότι ορισμένε εταιρείε θα ήθελαν. Το ερώτημα όμω είναι, διαφημίζει, διαφημίζει κανεί μια νέα ποικιλία και διαφημίζοντα την. Δηλαδή διαφημίζεται ότι έχει κάποια θρεπτικά υλικά ή αναφέρεται στην επισήμανση μονάχα ότι είναι ή δεν είναι GMO. Άρα επισήμανση για διαφήμιση είναι μια υπόθεση βεβαίως ξεχωριστή και ίσως θέλετε να δώσετε όσο περισσότερες, περισσότερη ενημέρωση θέλετε στους καταναλωτές. Αν θέλετε τώρα να τα επισημάνετε ως GMO, άλλη υπόθεση είναι βεβαίως. Ε. Η μας πεποίθηση είναι ότι οι τεχνικές αυτές, συνένεση εδώ των περισσότερων επιστημόνων, δεν είναι GMO, δεν είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και μπορούν να ωφελήσουν την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αν λάβουμε τώρα την εσφαλμένη απόφαση, θα πληρώσουμε το τίμημα αργότερα όλοι μας. Okay. Ο κύριος Χόισλινγκ, παρακαλώ. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν με ικανοποίησε η απάντηση της Κομισιόν. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένο. Βεβαίω έχει εμπιστοσύνη στην Κομισιόν, αλλά δεν μπορεί να την αφήσει μόνη τη στην υπόθεση αυτή. Ω Επιτροπή Γεωργία θα πρέπει να εξετάσουμε αν συμμετέχουμε και εμεί ω συναπόφαση δηλαδή ή αν ε, παίζουμε ένα δευτερεύοντα ρόλο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσει η νομική υπηρεσία της Επιτροπής Γεωργίας. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Στη Γερμανία διεξάγεται ήδη εδώ και καιρό συζήτηση για την ερμηνεία και βεβαίω γνωρίζω ότι η συζήτηση αυτή πολύ γρήγορα θα γίνει πολιτική συζήτηση και δεν επιτρέπεται να την παρατείνουμε και πάρα πολύ. Αλλά ούτε να δεχθούμε να μας παραμερίσουν διότι είναι σημαντικές οι συνέπειες των αποφάσεων αυτών. Και οι χώρες μέλη θα αρκεστούν να αφήσουν τα πράγματα στα χέρια της Κομισιόν ξαναλέω ότι ίσως η γραμματεία μπορεί να εγκύψει στο θέμα και να το συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ο κύριος Χαϊταμα. Να είμαι σύντομος. Πρέπει να προσέχουμε να μην φοβόμαστε τις νέες τεχνολογίες. Άκουσα μια φορά ότι ακόμα και κάποιες μη καπαό θέλουν να έχουν επισήμανση για προϊόντα που παράγονται χωρί βιοτεχνολογίε, ε, γιατί εκεί κάνουμε το αντίστροφο πρέπει να δούμε τι είναι ασφαλέ, τι είναι πολύ υποσχόμενο και τι προσφέρει δυνατότητε για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον κόσμο Όπω είπαμε σήμερα το ότι πρέπει να θρέψουμε περισσότερους αλλά με ε, τρόφιμα καλύτερη θρεπτική αξία, μειώνοντα ταυτόχρονα τι επιπτώσει για το περιβάλλον ε, για τι κλιματικέ αλλαγές κτλ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να κάνουμε τις σωστές επιλογές και σε καμία περίπτωση να μην ε, αμυνόμαστε κατά των τελευταίων τεχνολογιών αλλά να τις ε, ε, εντάξουμε στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Τώρα ολοκληρώσαμε και το δεύτερο γύρο. Ευχαριστούμε θερμά τους εμπειρογνώμονες καλεσμένους μας, γιατί σίγουρα με τις παρουσιάσεις τους εμπλούτησαν τη συζήτηση, μας τροφοδότησαν ε, με νέες πληροφορίες και νέα γνώση και πολλά θέματα θα πρέπει να διευκρινιστούν και περαιτέρω. Γιατί το ζήτημα είναι δύσκολο, περίπλοκο, ευαίσθητο για την κοινή γνώμη. Και είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις προκειμένου να θρέψουμε τον πλανήτη και στο μέλλον. Γιατί μέχρι το 2050 θα έχει πολλαπλασιαστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός. Αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε πιο ανοιχτοί και προς τις ε, νέες προπτικές Γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την παραγωγή μόνο των παραδοσιακών και συμβατικών ε, τρόπων καλλιέργειας. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους καλεσμένους και από τον πρώτο γύρο και από το δεύτερο γύρο της δημόσιας ακρόασης. Την ολοκληρώνουμε. Μια πολύ σύντομη τεχνική διακοπή και θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα, τη γνωμοδότηση του κυρίου Νταντά, που περιμένει ανυπόμονα. Ένα λεπτάκι μόνο διακοπή για να ξεπροβοδίσουμε τους καλεσμένους. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, πολιτική συνοχή στις ορεινές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάκτης γνωμοδότησής μας είναι ο κύριος Νταντά. Λάβαμε απόφαση να συντάξουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή Γεωργίας ε, επί της έκθεσης ε, πρωτοβουλίας μη νομοθετικού χαρακτήρα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης με θέμα την πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί στις περιοχές αυτές υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τη Γεωργία. Γι' αυτό λοιπόν κρίναμε σκόπιμο να συντάξουμε και εμείς γνωμοδότηση, την οποία αναθέσαμε στον κύριο Νταντάν. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο για να μας την παρουσιάσει. Παρακαλώ κύριε Νταντάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε πρόκειται για χθες πρωτοβουλία. Και εμείς πρέπει να δώσουμε μια γνωμοδότηση για την γεωργική πτυχή. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση, το κείμενο της οποίας είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Και εγώ είχα τη δυνατότητα να το συμπληρώσω στο σχέδιο γνωμοδότηση που έγραψα υπό τη μορφή τροπολογιών στην επόμενη φάση. Εγώ σα προτείνω, δεδομένων των ε, δικών μα ε, προβληματισμών και των εκθέσεων τη δική μα Επιτροπή επί του θέματο, και έχω στο νόμο ιδιαίτερα την εκθέση Dorfman για τα προβλήματα της ε, παραγωγής γαλακτός ε, σε ορεινές περιοχές να επιμείνουμε σε τρία κεφάλαια πιο συγκεκριμένα στα ζητήματα διακυβέρνησης και συνέργειας των ε, Ταμείων Συνοχής αφενός, στα ζητήματα επένδυσης ανταγωνιστικότητας και οικονομικής διαφοροποίησης, στις ορεινές περιοχές και τρίτον στην συγκεκριμένη ειδική διάρθρωση της ε, διατροφικής αλυσίδας στις ορεινές περιοχές όπου έχουμε μικρές εκμεταλλεύσεις, πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις που μεταποιούν στις παραγωγές τους και πολλά, ε, πολλά μικρά κυκλώματα. Ε, υπενθυμίζω στο σχέδιο γνωμοδοτησής μου ότι έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη ε, στον τομέα της συνοχής όταν μεταρρυθμίσαμε την ε, κοινή πολιτική γιατί τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος πυλώνας επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να στοχεύσουμε συγκεκριμένες πιστώσεις ε, για συγκεκριμένες περιοχές ε, όταν υπάρχουν φυσικοί περιορισμοί όπως οι ορεινές περιοχές λόγω, γιατί έχουμε τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά, την απομόνωση όλα αυτά αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες για αυτές τις περιοχές από οικονομική άποψη περιοχές αυτές, ε, στις διάφορες χώρες, ε, ε, καλούνται να δείξουν συνοχή στις διάφορες επιλογές για αυτές τις περιοχές. Σημειώνω, στον παροδότη, στη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει μια συγκεκριμένη παράγραφος που αφορά τις ορεινές περιοχές, τις νησιωτικές περιοχές και τις εξόχως απόμακρέ περιοχές. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε καμία πολιτική για τις ορεινές περιοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ε, με την ιδέα του να διαχωρίσουμε τις περιοχές αυτές σε ζώνες διότι οι ορεινές περιοχές ποικίλουν από χώρα σε χώρα οι χώρες είναι, οι είναι αυτές που ορίζουν ποιες είναι οι ορεινές περιοχές με κριτήρια τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε ορισμένες φορές είναι αρκετά διαφορετικά Αυτά ε, θα ακούσω με πολύ προσοχή ε, όσα έχουν να πούνε διάφοροι συνάδελφοι και θα λάβω υπόψη τις προτάσεις τροπολογιών ώστε η γνωμοδότησή μας να αντικατοπτρίζει με τον πιο πιστο δυνατό τρόπο τις εργασίες της δικής μας Επιτροπής. Σίγουρα υπάρχει επιτακτική ανάγκη να βοηθήσουμε στο μέλλον κυρίως αγροτικές εκμεταλλεύσεις ε, που βρίσκονται σε αντίξωες συνθήκες και κυρίως ε, στις ε, ορεινές περιοχές γιατί εκεί και η υποδομή είναι πιο δαπανηρή και το κόστος παραγωγής πιο υψηλό. Οπότε καλό θα ήταν ε, όλα αυτά που θα πούμε στην γνωμοδότησή να τα λάβουμε υπόψη και στη συζήτηση για τις προοπτικές της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2020. Το λόγο ζήτησε ο κύριος Ντόρφμαν. Όχι, η κυρία Σένερα. Η κυρία Σένερα. Πρώτα η κυρία Σένερα, μετά ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση κατά τη γνώμη μου και η έκθεση, γιατί όντως ε, οι ορεινές περιοχές δεν αντιχάνουν τους δέουσες προστασίας, ούτε λαμβάνουν ε, σημαντική βοήθεια και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται είτε από τα κράτη-μέλη είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ισπανία οι αυτονομίε είναι αρμόδιε. Ε, οι αρχές τη Γαλλική αποφασίζουν, τη αυτόνομη περιφέρεια. περιφέρειας. Και ε, παρατηρούμε το φαινόμενο της απερίμωση σε πολλές ορεινέ περιοχές. Ερωτώ λοιπόν, μήπως θα μπορούσαμε στην γνωμοδότηση να συμπεριλάβουμε και το θέμα των υπηρεσιών στι ορεινέ ε, περιοχέ. Παιδεία, υγεία, γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές οι υπηρεσίες ε, και η εξασφάλιση της παροχής τους για να παραμείνει ο πληθυσμός σε αυτές τις ζώνες. Γιατί είναι σημαντικό το θέμα της οικονομίας, η επιβίωση των εκμεταλλεύσεων, αλλά στη Γαλλικία και στην Ισπανία οι ορεινές ε, περιοχές εξαρτώνται κυρίως από την κτηνοτροφία, από την παραγωγή βόλιου κρέατος συγκεκριμένα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, αυτό το θέμα να το εξετάσουμε σφαιρικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριος ε, Ούτσεφ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι γιατί η γνωμοδότηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές περιοχές. Γιατί ήδη η κυνηγιορική πολιτική προβλέπει κάποια μέτρα για αυτές, αλλά και τα προγράμματα LIFE και ορίζοντας 2020 προβλέπω κάποια μέτρα. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε μία σφαιρική ε, συνολική προσέγγιση για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Και στις πιο φτωχές περιοχές ε, δεν έχουμε καν κατάλληλες υποδομές. Έχουμε απερίμωση, λίγες αρρώσιμες καλλιέργειες και υψηλότατο κόστος παραγωγής. Και αυτές ε, οι τάσεις χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Εκεί πάνω από το 60% των εδαφών της Βαλκανικής Χερσονήσου, για παράδειγμα, είναι ορεινές περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις ορεινές περιοχές να αναπτυχθούν περισσότερο και κυρίως ε, στη νότιο-ανατολική Ευρώπη όπως έγινε με τα Καρπάθια Όρη. Επίσης, ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία να αναπτυχθεί, να αναπτύξει τον τουρισμό της, αλλά και τη γεωργία της. Και καλό θα ήταν στην έκθεση να προσθέσουμε και άλλα σημεία. Για παράδειγμα, ε, το θέμα της ποιότητας ε, των ε, προϊόντων της ορεινής γεωργίας ή παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ή να δώσουμε κίνητρα σε νέους γεωργούς, ιδιαίτερα στις περιοχές αυτές. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, ο πρόεδρος. Ο κύριος Αντρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να εκφράσω τη συμφωνία μου για τη δημιουργία ζωνών με τον κύριο Νταντά. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ωστόσο αυτό το ζήτημα ε, Ξέρετε, έχουμε, έχει αυτή το πρόβλημα των φυσικών μειονεκτημάτων που ακούμε κάθε φορά που προτείνονται μεταρρυθμίσεις. Οι δύο πτυχές, ε, η γεωργική και ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ορεινών ζωνών. Όσον αφορά τη γεωργική πτυχή, ε, όταν μιλάμε για φυσικά μειονεκτήματα, κατά την απόψή μου, πρέπει να βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες των περιοχών και τη δική μας πολιτική βούληση. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ένα βασικό βήμα στον πρώτο πυλώνα. Αυτή είναι η απόψη μου. Όσον αφορά την ανάπτυξη τη υπαίθρου, επειδή ακριβώ στι περιοχέ αυτέ υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα απομάκρυση υψομέτρου, κλίματο, προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε, πιστεύω ότι εκεί πρέπει να υπάρχουν διαφορετικέ προποθέσει ε, παροχή βοήθεια ώστε να βοηθάμε με ίσο τρόπο όλες αυτές τις περιοχές, με ισχυρό τρόπο και σαφή τρόπο σε σχέση με τις άλλες περιοχές των ε, κρατών μελών και τις αστικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω ότι αυτή η εκθέση θα πρέπει να αποτελεί αφετηρία για να ξεκινήσει ένας πραγματικός προβληματισμός όσον αφορά τις ε, ε, ειδικέ ε, δημόσιες πολιτικές για αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές όπως οι ορεινές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή έχει θεμελιώδη σημασία. Μια και οι χώρες που λαμβάνουν τα Ταμεία Συνοχής, οι δικαιούχοι των κονδυλίων της Συνοχής, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μάλιστα και οι περιοχές που λαμβάνουν τέτοια κονδύλια συνοχής έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, συγκρίσιμα. Οι ορεινές περιοχές έχουν μια οικονομία που προσπαθεί να εξασφαλίσει την ευημερία του πληθυσμού, υπό αντίξεως όμως συνθήκες. Πολύ συχνά η παραγωγή στις ορεινές αυτές περιοχές παράγουν τα ίδια προϊόντα που, με τους παραγούς της παιδιάδας για παράδειγμα, αλλά με πολύ ψηλότερο κόστος παραγωγής. Οπότε έχουν χαμηλότερα εισοδήματα, με αποτέλεσμα η απασχόληση να χωλαίνει. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε τη γεωργία και την παραγωγή στις ορεινές περιοχές. Ένα τμήμα των προβλημάτων θα το λύσουμε με τις επενδύσεις αλλά και τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Ως και ηγητής στη γνωμοδότηση αυτή και ως νέος ευρωβουλευτής θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό και Χρειαζόμαστε και μέσα επικοινωνίας και μέσα συγκοινωνίας, καλύτερες υποδομές και ίσες ευκαιρίες για όλους. Παρόμοια πρόσβαση και στο ευρυζωνικό ίντερνετ. Και για να επανέλθω στην πρόταση του κυρίου Ρούτσεφ, καλό θα ήταν να έχουμε και ένα σήμα ποιότητας για τα προϊόντα της ορεινής γεωργίας, για να τα προωθήσουμε περισσότερο. Γιατί υπάρχει σήμα για τα τοπικά προϊόντα, αλλά δεν τα έχουμε αξιοποιήσει αρκετά. Θα συνεργαστώ με τον κύριο Νταντάν πάντως για να εμπλουτίσουμε την γνωμοδότησή του. Η κυρία Γκιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω και εγώ κάποια σχόλια και κάποιες ιδέες για την έκθεση. Υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ εύστοχο το επισήμανε ο κύριος Νταντά. Το πρώτο πρόβλημα αφορά την λήψη υπόψη των ορεινών περιοχών στα κράτη-μέλη και δεν είναι καθόλου εύκολο να το επιλύσουμε. Γιατί κάθε χώρα διαφορετικά αντιμετωπίζει τις ορεινές περιοχές και τις δυσκολίες τους. Καλό θα είναι υπάρχει μια σύγκληση όμως στο θέμα του πώς ορίζουμε τις ορεινές περιοχές και πώς αντιμετωπίζουμε. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και τα προβλήματά τους αν έχουμε πιο εναρμονισμένη προσέγγιση. Αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο. Επίσης είπατε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι βασικές υπηρεσίες. Αλλά όλη η πολιτική συνοχής και στην Ήπεθρο και στις ορεινές περιοχές αν δεν προβλέπει χρηματοδότηση των υποδομών και των βασικών υπηρεσιών ουσιαστικά θα φέρνει τις περιοχές αυτές σε δυσμενή θέση σχέση με τις υπόλοιπες. Οπότε η συνοχή θα εξασφαλιστεί με την εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών. Γιατί εκτός του φυσικού μειονεκτήματος και της απόστασης ή της ε, δύσκολη προσπέλασης, καλό θα ήταν τουλάχιστον να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στι υποδομέ παρόμοια με την υπολείπων περιοχών. Επίσης, γεωργία και προϊόντα. Για να μειωθεί το κόστος παραγωγής θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση στις υποδομές και να δοθούν κίνητρα για τους νέους. Γιατί αλλιώς πώς θα πάνε να ζήσουν οι νέοι σε περιοχές ε, που θα θεωρήσουν ότι είναι μειονεκτικές και για το μέλλον τους. Θα καταθέσω τροπολογίες λοιπόν για την γνωμοδότηση, γιατί και στις ορεινές περιοχές, όπως ισχύει γενικά στην Ήπεθρο, έχουμε πολλαπλές δραστηριότητες και έτσι συγκροτείται το εισόδημα. Κάποιος έχει μία μικρή ε, εκμετάλλευση, ταυτόχρονα τη χρησιμοποιεί και για αγροτουρισμό γίνεται ένα συνδυασμό των δραστηριοτήτων. Αυτό συμβαίνει στην Ισπανία, φαντάζομαι θα συμβαίνει και αλλού, αλλά πολλές φορές δημιουργεί πρόβλημα αυτή η πολλαπλή δραστηριότητα και το πώς λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του εισοδήματος. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια ιδέα, μια έννοια της οικογενειακής εκμετάλλευσης, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε συμπληρωματικότητα του εισοδήματος από διάφορους οικονομικούς τομείς. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τις ορεινές περιοχές, ισχύει γενικώ για την Ήπεθρο. Να λάβουμε υπόψη λοιπόν τις οικογενειακές επιχειρήσεις που θα συμπληρώνουν αυτή την πολλαπλή δραστηριότητα. Έτσι θα δώσουμε κίνητρα και σε νέους και στον κόσμο να πηγαίνει για να ζήσει, να σε τέτοιες περιοχές ορεινές. Θα πρέπει η κοινή γεωργική πολιτική να λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών. Στη, σε εμάς ε, υπάρχει πρόβλημα με τον ε, συντελεστή της ε, επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων. Γιατί μερικές ζώνες έχουν ιδιαιτερότητες και δεν λαμβάνονται αυτές υπόψη πάντα στην κοινή γεωρική πολιτική. Έρχεται η κοινή γεωρική πολιτική και με τους συντελεστές που επιβάλλει διακόπτει την ε, σωστή προστασία συγκεκριμένων ζωνών. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για αγροτικές ζώνες με φυσικά μειονεκτήματα. Εκεί θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και να αναγνωρίσουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες στην κοινή γεωργική πολιτική. Επαναλαμβάνω, θα καταθέσω και τροπολογίες ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση όπως θέλει και ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάναγκαν. Uh, uh, Σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικός ο τομέας αυτός και οφείλω να ομολογήσω ότι με απογοητεύει η περιορισμένη παρουσία βουλευτών. Πώς κατεβαίνουν στις εκλογές και μετά ε, δεν έρχονται εδώ να εκπροσωπούν τους ψηφοφόρους. Ορισμένοι θα πούνε ότι είναι αργά το βράδυ. Να το πείτε στον πατέρα μου που δουλεύει, είναι 70 χρονών και εξακολουθεί δουλεύει, να δουλεύει και μέχρι, θα δουλεύει μέχρι το βράδυ. Να τα πείτε αυτά και στου αντιπάλου τη Ευρώπη ή του ευρωσκεπτικιστέ, όπω εγώ και ο γείτονά μου πίσω, και οι άλλοι που θέλουν να διοικοτομήσουν την Ευρώπη που είναι. Άνθρωποι που δουλεύουν αγρότε σε, αυτές, σε αυτού του τομεί, προσφέρουν περιβαλλοντικέ υπηρεσίε, τουριστικέ υπηρεσίε, βεβαίω τρόφιμα, παράγουν τρόφιμα, ε, διαχείριζουν το περιβάλλον και στην Ιρλανδία τουλάχιστον σε πολλές από τις περιοχές αυτές και στους τονείς αυτούς κρατάνε και σε ζωή την ε, Ιρλανδική γλώσσα. Υπάρχουν ιστορικοί λόγοι. Υπάρχουν ιστορικοί λόγοι για τους οποίου διατηρήθηκε εκεί, στα δύσβατα αυτά εδάφη, η Ιρλανδική γλώσσα, γιατί εκεί κατέφευγαν. Διατηρείται όμω ζωντανή και αυτή εδώ η έκθεση είναι σημαντική τις τελευταίες μέρες συνομιλούσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περιοχή αυτή γενικότερα. Αν θέλουμε να σεβαστούμε και πραγματικά αν ενδιαφερόμαστε για τους αγρότες αυτών των δύσκολων περιοχών πρέπει να ξεχάσουμε επιτέλους ότι είναι αυτοί οι οποίοι είναι τελευταίοι που πληρώνονται και όταν πάτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάτε και τους ρωτήσετε γιατί είμαστε τελευταίοι που μας πληρώνετε. Είστε τελευταίοι από ολόκληρη την Ευρώπη που πληρώνονται, μας απαντούν τότε. Εμείς σεβόμαστε τις περιοχές αυτές. Δεν θα πρέπει να είναι οι τελευταίοι που πληρώνονται, ούτε να έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες μέχρι ότου να πληρωθούν. Και για την Ιρλανδία τουλάχιστον έχουμε μια καταπληκτική κατάσταση όπου ο κόσμος που ζει στην Ήπεθρο που δύσκολα τα βγάζουν πέρα λαμβάνουν τελικά τις μικρότερες πληρωμές. Ακόμα και στον πυλώνα 2 όπου ίσως είχαν κάποια ελπίδα να πάρουν κάποια χρήματα φαίνεται ότι θα τους αναγκάσουν να ξεπεράσουν τόσα πολλά εμπόδια που ακόμα και τότε θα φτάσουν σε μεγάλη απόσταση από τον πιο εύπορο αγρότη που παράγει δημητριακά. Αν θέλουμε λοιπόν να σεβαστούμε τις περιοχές αυτές πρέπει να τις πάρουμε σοβαρά υπόψη και να μην δυσκολεύουμε τον κόσμο που ζει σε αυτές. Όταν συναντήθηκα με εκπροσώπους της Κομισιόν τους μίλησα για την ιδέα αυτή ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μειονεκτικοί μειονεκτούν δηλαδή οικονομικά, γιατί υπάρχουν και πολλοί περιορισμοί για τις γέες αυτές. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την οδηγία Habitat ή άλλες σχετικές. Πρόβλημα έχω με το γεγονός ότι ο κόσμος τελικώς μειονεκτεί, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση οικονομικά λόγω αυτών των περιορισμών. Και ούτε μπορείτε, μου είπε η Κομισιόν, να αναμένετε ότι θα σας αποζημιώσουμε 100%. Γιατί όχι όμως γιατί όχι, θυσιάζουν κάποια πράγματα να έχουν οικονομική αντιστάθμιση. Ούτε μου είπαν μπορείτε να αναμένετε να σας πληρώνουμε για πάντα. Μα ναι, οι περιορισμοί θα υπάρχουν όμως για πάντα. Αν υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί στη διαβίωση των ανθρώπων αυτών εκεί επί τόπου, για πάντα, αν θέλετε πραγματικά να αποδώσετε κάποια αξία, γιατί αξία σημαίνει βάζεις και ένα τίμημα. Γιατί αλλιώ θα καταλήξετε σε μια κατάσταση που θα εγκαταλείψουν τις γέες αυτές. Και πολλές, πολλά από, τα, πολλές από τις περιοχές αυτές είναι περιοχές όπου το τοπίο το διαχειρίζονται οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Πολλοί από αυτούς θέλουν να συνεργαστούν και θέλουν να πετύχει η υπόθεση αυτή. Εγώ πήγα σε μια συνάντηση με πολλούς προβατοτρόφους και μερικοί είπαν ότι θέλουν να φέρουν τον αητό στις περιοχές του και αντί να τον ε, ε, επιτιμήσουν οι υπόλοιποι, τελικά τον επεφήμισαν οι υπόλοιποι. Αυτοί όμως την πατάνε τελικά όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα. Αυτούς θα τους πληρώνετε πρώτους, όχι τελευταίους. Αυτή είναι η κατάσταση στην πατρίδα μου. Στην πατρίδα μου έχουμε πολλά προβλήματα. Πληρώνουμε τους επικεφαλείς ορισμένων αγροτικών σωματείων ένα μισό εκατομμύριο το χρόνο. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πράγματι συμφωνώ για τη σπουδαιότητα αυτής της έκθεσης ε, λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά ένα ενιαίο έδαφος όπου αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες όλοι οι αγρότες όσον αφορά την παραγωγή ούτε επιτυχάνουν τα ίδια αποτελέσματα. Ε, ο συναδελφός μου από τη δυτική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις μίλησε και εγώ τώρα θέλω να σας παρουσιάσω ότι συμβαίνει στην ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, σε κάθε χώρα οι συνθήκες ε, γεωργικής παραγωγής είναι διαφορετικές. Το ερώτημα είναι πώς ε, εξομοιώνουμε όλα αυτά, πώς αντισταθμίζουμε τα προβλήματα. Για παράδειγμα στη Λιθουανία, δυστυχώς πρέπει να παραδεχτώ ότι για την περίοδο 2014-2020 δεν υπάρχει κανένας χάρτης που να καθορίζει τις περιοχές ε, που δεν είναι τόσο κατάλληλες για γεωργική παραγωγή. Θεωρείται δηλαδή ότι όλα τα εδάφη στη Λιθουανία είναι ευνοϊκά για τις καλλιέργειες, το οποίο δεν είναι αληθές και φυσικά ορισμένοι γεωργοί που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες δεν πρόκειται να λάβουν κάποια αποζημίωση. Εγώ ίδιος προέρχομαι από μια περιοχή κοντά στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περιοχή αυτή δεν είναι τόσο δημοφιλής, ούτε πολυπληθής. Ο κόσμος φεύγει από την περιοχή αυτή. Ε, η περιοχή που ζω βρίσκεται επίσης πολύ κοντά σε, ένα πυρηνικό εργοστάσιο όπου υπάρχει και μια προστατευόμενη περιοχή όπως υπάρχουν γύρω από τα πυρηνικά εργοστάσια. Οι άνθρωποι ξέρετε τείνουν να φεύγουν από αυτές τις περιοχές, δεν θέλουν να τις καλλιεργήσουν, δεν είναι βέβαιο ότι είναι ασφαλείς υπάρχει ε, μια δυσχέρεια, μια δυσπιστία προς τη ζωή σε αυτές τις περιοχές. Επίσης υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα που αφορά τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Λόγω των χαμηλών ε, εισοδημάτων οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις αγροτικές δραστηριότητε και πηγαίνουν να αναζητήσουν την τύχη τους ε, στην Δυτική Ευρώπη, στις βόρειες χώρες, στις σκανδιναβικές χώρες, στην Ισπανία, στη Γερμανία. Στη Λουθανία, για παράδειγμα, έχει φύγει το 1 τέταρτο του πληθυσμού σε ηλικία εργασία εντό 15 ετών. Είναι μεγάλο το αυτό το πρόβλημα. Φυσικά οι άνθρωποι που ζουν φυσιολογικά ε, έχουν τις ίδιες δραστηριότητες, ε, ε, εκτρέφουν πρόβατα, έχουν καλλιέργειες, ε, και θα έμεναν οι άνθρωποι φυσικά στη χώρα να ανταμείβονταν καλύτερα με τρόπο ανταγωνιστικό προς τις ε, δυτικές χώρες. Του χρόνου θα αξιοποιήσουμε την επιτυχία της, θα αξιολογήσουμε την ε, επιτυχία της νέας γεωργικής πολιτικής και κατά πόσο συνέβαλε στην ανανέωση, στην αναζωογόνηση ουσιαστικά της γεωργίας και στη διατήρηση των ανθρώπων στις γεωργικές δραστηριότητες εκεί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα προβλήματα που ανέφερα εγώ και πιστεύω σε αυτήν την έκθεση ε, αποτυπώνονται εν μέρη τα προβλήματα γιατί μιλάμε για τις ορεινές περιοχές αλλά ε, θα πρέπει επίσης να δούμε όλες τις ε, μειονεκτούσες περιοχές όχι μόνο τις ορεινές οι αποζημιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αποτελούν απλά πηγή κέρδους. Πρέπει να είναι ένας αντισταθμιστικός μηχανισμός που να θέτει όλους τους γεωργούς ε, λίγο πολύ τις ίδιες συνθήκες ε, χωρίς να χρειάζεται αυτοί να ε, μεταναστεύουν αναζητώντας καλύτερη τύχη. Ευχαριστώ. Ντόρφμαν. Ο κύριο Νταντέν συνέταξε μια σημαντική έκθεση και τον ευχαριστώ. Όπως είπαν και άλλοι πριν, αυτές οι ορεινές περιοχές είτε θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο μιας ιδιαίτερης πολιτικής, είτε θα δούμε να πεθαίνουν αργά, αλλά σίγουρα. Και αν δεν το πιστεύετε, μπορείτε να πάτε να δείτε σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, εκεί στην ε, Βόρεια Ιταλία, στο Τυρόλο, στην Μπερνίνα, μπορείτε να δείτε τι γίνεται. Έχουν νεκρώσει περιοχές ολόκληρες. Εάν δεν φτιάξουμε μια πραγματική πολιτική για τις ορεινές περιοχές δεν θα λειτουργήσει. Αυτά που λένε οι επίτροποι ότι υπάρχουν τα εργαλεία στην ε, περιφερειακή πολιτική που επιτρέπουν να ε, δημιουργηθούν τις πολιτικές. Μπορεί να είναι σωστό αυτό, αλλά ποιες χώρες τα πράττουν αυτά. Για την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, όλα αυτά είναι περιθώριο δεν έχουν κανένα πραγματικό ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται αλλού. Για παράδειγμα, γαλακτοπαραγωγή, μέγα πρόβλημα. Η γαλακτοπαραγωγή στα βουνά δεν τα καταφέρνουν να επιβιώσουν. Και πάμε να φτιάξουμε ένα ιδιαίτερο ταμείο για τη γαλακτοπαραγωγή με 500 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουν υποστήριξη στο, στην παραγόμενη ποσότητα. Όποιος παράγει πολύ, όποιος παράγει μεγάλη ποσότητα, παίρνει πολλά χρήματα. Όποιος παράγει μικρές ποσότητες, παίρνει λίγα. Έτσι δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Σας λέω ένα παράδειγμα. Όταν τώρα στους κάμπους υπάρχει μια, ε, γίνει μια πλημμύρα, τότε λέμε όλοι «Α, αυτή η αλλαγή του κλίματος». Δέστε τις μεγάλες πλημμύρες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και συγκρίνεται τις τη βροχοπτώσεις και θα δείτε τελικά ότι δεν έχουν πολύ σχέση με την αλλαγή του κλίματος. Το πρόβλημα είναι ότι πέφτει η βροχή στα ορεινά και καταλήγει ταχύτατα στις κοιλάδες διότι έχει διαβρωθεί το έδαφος στα ορεινά επειδή κανείς δεν είναι εκεί να τα φροντίσει. Και έτσι έρχεται ολόκληρη η αλυσίδα των επιπτώσεων. Επειδή δεν υπάρχουν πλέον άνθρωποι στα βουνά για να φροντίζουν το περιβάλλον. Πρέπει να εξασφαλιστεί το εισόδημα των ορεινών πληθυσμών και χρειάζεται ειδική πολιτική γι' αυτό. Ούτε νομίζω θα κοστίσει και πάρα πολλά. Χρειάζεται ωστόσο μια ορθή και ορθολογική προσέγγιση. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ντούμητρου. Thank you very much, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ανταλλάξουμε απόψη επ' ευκαιρία αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας και σας διαβεβαιώ ότι είμαστε πρόθυμοι ε, για οποιαδήποτε ενημέρωση και διευκρίνηση για θέματα πολιτικής συνοχής στις ορεινές περιοχές. Οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 20% περίπου της ε, ευρωπαϊκής επικράτειας και χαρακτηρίζονται από μεγάλη εδαφική και κοινωνική ποικιλομορφία. Έχουμε ήδη μακρά ιστορία στην κυνηγιορική πολιτική που δίνει σημασία ιδιαίτερη στις ορεινές περιοχές. Και μάλιστα ένα σταθερό στοιχείο είναι ο ορισμός των ε, ορεινών περιοχών. Έχουμε στην ε, περιφερειακή πολιτική ορισμό που λαμβάνει υπόψη το υψόμετρο, την κλίση. Έχουμε συγκεκριμένο ορισμό που δεν έχει αλλάξει από την αρχή. Και μάλιστα με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αλλάξαμε μερικές φορές τα κριτήρια ε, χαρακτηρισμού ορισμένων περιοχών, αλλά αυτό δεν ισχύει για τις ορεινές περιοχές, για τις οποίες ο ορισμός είναι ο ίδιος από παλιά. Οπότε αναγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες, ε, δύσκολη τοπογραφία, απομακρυσμένες περιοχές, αντίξουες ε, κλιματικές συνθήκες. Αυτές είναι μερικές από τις αντικσότητες και τις ιδιαιτερότητες αλλά έχουμε και κάποια ατού, το μοναδικό τοπίο, την βιοπικιλότητα, ε, υδροφόρους ορίζοντες, πολιτιστική παράδοση. Πολλά προτερήματα και για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών που μπορούν να απτύξουν τον αγροτουρισμό. Και εγώ κατάγομαι από ένα χωριό της Ρουμανίας ε, ορεινό και γνωρίζω την αλληλεγγύη μεταξύ των ορεσιβίων. Επίσης ε, αναγνωρίζουμε στην κοινή γεωρική πολιτική το ρόλο και τη σημασία των ορεινών περιοχών και έχουμε προβλέψει πολλούς μηχανισμούς για τη στήριξή τους. Ήδη υπάρχει η δυνατότητα στήριξης των ορεινών περιοχών για να επιβιώσουν οι γεωρικές δραστηριότητες και εκεί. Και όλοι αναφερθήκατε στις δυσκολίες που έχουν οι ορεινές περιοχές. Ε, έχουμε δυνατότητα καταβολής αντισταθμιστικών πληρωμών για να διατηρηθεί η γεωρική δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές. Και αυτό είναι επιπλέον του εισοδήματος και παντού μπορεί να δοθεί αντιστάθμιση στους γεωργούς που ζητούν τέτοιες αντισταθμιστικές πληρωμές. Και μάλιστα ε, αυτό γίνεται συνεχώς. Όσο υπάρχει ζήτηση αυτά τα προγράμματα παρέχουν τέτοια δυνατότητα. Αυτές οι αποζημιώσεις αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα αυτών των περιοχών, υπερβολικό κόστος παραγωγής και χαμηλότερο εισόδημα. Και υπάρχουν κατώτατα και ανώτατα όρια στην νομοθεσία. Το μέγιστο όριο είναι ανώτερο μάλιστα από αυτό που πληρώνουμε ε, σε άλλες περιοχές με ε, φυσικά μειονεκτήματα. Και μέχρι στιγμής τα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν καλά τις ανάγκες ε, των ε, ορεινών περιοχών και την αντιστάθμιση των προβλημάτων. Σε 17 χώρες ε, υπάρχουν σχετικά προγράμματα και καλύπτουν 13 εκατομμύρια εκτάρια ορεινών εκτάσεων. Επίσης υπάρχει δυνατότητα με τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα για χορήγηση αντισταθμιστικών πληρωμών για τους αγρότες ορεινών περιοχών ή περιοχών με άλλους φυσικούς περιορισμούς. Τώρα, για τη Λιθουανία. Η Λιθουανία δεν έχει βουνά σε σχέση με τον ορισμό, αλλά μπορούμε, μπορούμε να προβλέψουμε τις εθνιστικές πληρωμές για τις περιοχές που έχουν άλλου είδους φυσικούς περιορισμούς. Δεν εμπίπτουν όμως τις ορεινές. Πάντως οι αντισταθμιστικές πληρωμές είναι η σημαντικότερη παρέμβαση που μας επιτρέπει η κοινή γεωργική πολιτική πέρα αυτών των περιοχών. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα για τη στήριξη των γεωργικών και άλλων δραστηριοτήτων στις ορεινές ζώνες. Ένα άλλο μέτρο που είναι πολύ σημαντικό είναι η πρακτική διαχείρισης ε, ακροπεριβαλλοντικού χαρακτήρα η εξασφάλιση υπηρεσιών για τη σωστή διαχείριση των πόρων και τη διαφύλαξη της βιοπικιλότητας και της υψηλής ε, αξίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. Ένα μεγάλο τμήμα των ε, ορεινών περιοχών καλύπτονται από δάση και από αλπικούς βοσκοτόπους. Για τα δάση έχουμε μια γκάμα μέτρων στήριξης. Αναδάσωση, πυρασφάλεια, και επενδύσεις για να εξασφαλιστεί πρόσβαση στα δάση και επένδυση σε δασικούς δρόμους. Και υπάρχουν δυνατότητες που ισχύουν γενικώ για την Ήπεθρο, με επιπλέον πλεονεκτήματα ή προνομιακή μεταχείριση για τις ορεινές περιοχές. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις ε, στις ορεινές περιοχές σε υποδομές έχουν υψηλότερο ε, ποσοστό στήριξης από ό,τι αντίστοιχε επενδύσει σε άλλες περιοχές με φυσικούς περιορισμούς. Και το πρόγραμμα Leader δίνει δυνατότητα. Το Leader καλύπτει και εδάφη σε ορεινέ περιοχές. Εκεί καλύπτονται ανάγκες συμπληρωματικών υποδομών. Και έχουμε και τα προγράμματα ανάπτυξης πέθρου που μπορούν να ωφελήσουν και ορεινές περιοχές. Επίσης μπορούμε να στηρίξουμε κάποιες ε, δραστηριότητες συνεργασίας ε, και την εταιρική σχέση για την καινοτομία. Τέτοια, τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να εφαρμοστούν και στις ορεινές περιοχές. Επίσης, οι ε, παραγωγοί στις ορεινές περιοχές μπορούν να, θέσουν σε εμπορία τα προϊόντα τους με ειδικό σήμα, ειδική έμφαση στον ορεινό τους χαρακτήρα, που δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και εμείς έχουμε έναν επιπλέον όρο ποιότητας, το ορεινό προϊόν. Έτσι οι ορινές περιοχές μπορούν να διαφημίσουν καλύτερα και να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις δυνατότητες που έχουμε μέσω της, των πολιτικών ανάπτυξη υπαίθρου να στηρίξουμε τις ορεινές περιοχές. Και φυσικά συμμετέχουμε και σε γενικότερες πρωτοβουλίες. Συνεργαζόμαστε με την Μοντάνα. Ε, συμμετέχουμε στην Σύμβαση για τις Αλπικές Ζώνες και έχουμε και την ε, μακροπεριφερειακή πολιτική για τις αλπικές περιοχές. Επίσης έχουμε και 250 μέλη στο πάνελ του ΟΗΕ για τις ορεινές περιοχές. Μάλιστα και οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση για τις Περιφέρειες μπορεί να προσθέσει κάτι αν θέλει. Η δική μας Γενική Διεύθυνση της Γεωργίας είναι πρόθυμη για συνεργασία με τον εισηγητή σας για παροχή πληροφοριών, γιατί έχουμε πολλές πληροφορίες για σχετικά πρόσφατα προγράμματα, τα οποία έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα καθέναν από τους ομιλητές για την συμμετοχή τους. Όλα αυτά μου φαίνεται ότι είναι πολύ λογικά. Η πρώτη ανησυχία πιστεύω των κατοίκων των ορεινών περιοχών είναι τα βουνά να μην θεωρούνται ένα μέρος όπου ε, προστατεύουμε κάποιους ε, ε, ντόπιου, ε, ηθαγενεί. Ε, θέλουν να του βλέπουμε σε αν περιοχέ με ειδικέ ανάγκε που χρήζουν προστασία. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, με την αντιστάθμιση. Πρέπει να προσέχουμε γιατί οι ενισχύσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε έναν συναγωνισμό στρεμάτο, στρεματικό. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης, της στρεματικής ενίσχυσης και μετά της αξιολόγησης της γεωργικής οικονομίας επιτόπου. Εκεί είναι, έγκυται όλες οι δυσκολίες και η κυρία Αγγιλέρα το είπε πολύ σωστά στη, λόγω της εποχικότητας το, ε, είναι δύσκολο να έχει κανείς μόνο μία δουλειά σε μια ορεινή περιοχή. Συνήθως οι άνθρωποι κάνουν πολλές δουλειές ε, όπου δεν δέχονται η μία την άλλη ή αλληλεπικαλύπτονται. Όταν μιλάμε λοιπόν για ορεινές περιοχές πρέπει να μιλάμε για γεωργούς αλλά ε, πρέπει να μιλάμε για εργαζόμενους γενικότερα, γιατί κάποιος μπορεί να είναι γεωργός, μια άλλη εποχή μπορεί να είναι καθηγητισκή, Πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη ε, αυτές τις πολλαπλές δραστηριότητες που εξαρτώνται από τις εποχές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ε, ε, θα, έτσι λοιπόν θα συνεχίσουν να ζουν να ζωντανά τα βουνά, να δώσουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους τους να αξιοποιήσουν όλους τους υπάρχοντες πόρους και όχι απλά να εντάξουμε τις ορεινές περιοχές να τις προσαρτήσουμε σε άλλες πολιτικές. Ε, οι πολιτικές για τα ισορρινές περιοχές πρέπει να είναι αυτόνομες ε, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών. Με εξαίρεση ως του leader που περιλαμβάνει αυτή τη διάσταση θα πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε οι ορεινές περιοχές να λαμβάνονται υπόψη ως ε, εδάφη και να έχουμε τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές. Σας ευχαριστώ. Στις 11 Ιανουαρίου θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, μέχρι 15 Ιανουαρίου έχετε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στις 23 Φεβρουαρίου. Περνάμε στο τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη, ε, ουσιαστικό, την ανταλλαγή απόψε με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για τη θέση σε ισχύ του κανονισμού για την πρόθεση. Στις αρχές του 2014 η κυρία Γκαρσία πραγματοποίησε άθλο πραγματικό, καταλήγοντας σε συμφωνία με το Συμβούλιο σε λιγότερο από ένα μήνα με δύο μόνο τριμέρες διαλόγους. Τώρα θα έχουμε παρουσίαση του κανονισμού αυτού για την πρόθεση από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιστροπής, τον κύριο Διέκο Κάνκαφάνο που θα μας ενημερώσει για το πώς πάει αυτός ο κανονισμός. Παρακαλώ κύριε Καγκαφάνο. Ευχαριστώ. Έχω τα, τις σημειώσεις μου στα αγγλικά, αλλά θα μιλήσω ισπανικά παρόλα αυτά. Ο κανονισμός ε, τίθεται σε ισχύ σήμερα. Γι' αυτό και σας ζήτησα να έρθω σήμερα για να σας τον παρουσιάσω, γιατί εξηγήσαμε σε πολλά κρατημέλη ότι ο κανονισμός αυτός βρήθη ευκαιριών αλλά τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής ε, ήταν υπεύθυνα, γι' αυτό κρίνομαι σκόπιμο σήμερα την ημέρα σε ισχύ του κανονισμού να σας τον εξηγήσω. Θα τα πω γρήγορα γιατί είναι ήδη αργά και είχατε και φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα. Το βασικό είναι ότι οι γραπιστιστικέ εξαγωγέ πάνε πολύ καλά. Καλύτερα από ποτέ, μάλιστα, θα έλεγα. Ποτέ δεν είχαμε τόσο σημαντικέ εξαγωγέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν ε, δείτε την κόκκινη γραμμή βλέπετε τι εξαγωγές έχουμε φέτος. Κάτι που μάθαμε όμως χάρη στο ρωσικό εμπάργο ή εξαιτία του είναι ότι θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις εξαγωγές μας, τους προορισμούς. Και ο κανονισμό αυτό που σήμερα μπαίνει σε ισχύ επιτρέπει ακριβώ τη διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Αυτό το κάναμε και στο παρελθόν. Εγκρίναμε πολλά προγράμματα και οι χώρε που ευνοήθηκαν κυρίω ήταν Ιταλία, Ελλάδα, από πολλά προγράμματα ε, ε, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία και μάλιστα θα ήθελα οι βουλευτές από χώρες που δεν ανέφερα να ε, παροτρύνουν τους οργανώσεις τους να υποβάλουν αιτήσει για χρηματοδότηση. Και τα προϊόντα που υποφελήθηκαν ήταν προκεφητικά, γαλακτοκομικά, ε, προέλευση, ονομασίες προέλευσης, βιολογική γεωργία και κρασί. Θα θέλαμε και στο μέλλον να, να χρηματοδοτήσουμε την προώθηση των προϊόντων αυτών και εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραλαμβάνω ο κανονισμό ε, τίθεται σήμερα σε ισχύ και είστε και πρωταγωνιστές ε, γιατί τον εγκρίνατε πέρυσι και ήδη έχουν εγκριθεί όλε οι κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικέ πράξει, γιατί πολλέ φορέ δημιουργούν προβλήματα οι πράξει αυτέ για την Επιτροπή Γεωργία. αλλά στην περίπτωση αυτή δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, Όλε εγκρίθηκαν, όλε δημοσιεύθηκαν και με τη συμφωνία τη Επιτροπή σα και όπω σα είπα ο κανονισμό μπαίνει σε εφαρμογή σήμερα. Σε αυτή τη διαφάνεια θα σταθώ λίγο περισσότερο γιατί περιλαμβάνει τις ε, καινοτομίες, τα νέα στοιχεία του κανονισμού αριστερά βλέπουμε ότι θέλουμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία στις εξαγωγές και έχουμε ετήσιο πρόγραμμα, θα σας το αναλύσω κατόπιν. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην πρόθεση, στρατής πρόθεση σε τρίτες χώρες, όχι μόνο στη δική μας αγορά. Θέλουμε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα και πολλά προγράμματα έχουν υποβληθεί από ιδιωτικό τομέα των χωρών και μάλιστα το ποστό χρηματοδότηση είναι πολύ πιο γενναιόδωρο ε, τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Ο νέος κανονισμός επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή και σε νέους δικαιούχους. Μπορούμε να συγχρηματοδοτούμε πολύ περισσότερα προϊόντα. Διαβρύθηκε και το πεδίο εφαρμογή των προϊόντων. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα σήματα, τα εμπορικά σήματα και την προέλευση. Έχουμε περισσότερα χρήματα και κονδύλια σε περίπτωση κρίση και θα συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα. Πάει ο ρόλος των κρατών μελών, θα σταματήσει η εθνική συγχρηματοδότηση. Θα έχουμε πιο απλούστατη, απλούστερη διαδικασία γιατί θα μας βοηθήσει και ο οργανισμός στο Λουξεμβούργο και το χαρμόσυνο μαντάτο είναι ότι έχουμε περισσότερα χρήματα, 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όπως είπα και προηγουμένως, ο νέος κανονισμός έχει έναν εταιρισμό. Χρηματοδοτεί πολύ περισσότερα προϊόντα, όλα τα γεωργικά πλην του καπνού Επίσης μπορούμε να συγχρηματοδοτούμε και με τα ποιημένα προϊόντα, σοκολάτα, μπύρα, ζυμαρικά και ε, θα δώσουμε ιδιαίτερα έμφαση στις γεωγραφικές ενδείξεις, ε, ονομασίες προέλευσης. Ε, για το κρασί έχουμε απλά προγράμματα και πολλαπλά προγράμματα εκεί που θα συνδυάζεται με άλλα προϊόντα και που θα είναι μόνο του. Επίσης ε, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και ευνοϊκή μεταχείριση για τις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές, για τα βιολογικά προϊόντα και για τις γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης. Ποιο μπορεί να υποβάλει αίτηση. Έχουμε διευρύνει και το πεδίο εφαρμογή των δικαιούχων, οργανώσει που εκπροσωπούν τον κλάδο είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οργανώσει παραγωγών, ακόμη και ε, σώμα, ε, οργανισμοί του δημόσιου τομέα. αυτή η αριστερή διαφάνεια θα ικανοποιήσει τον κύριο Ντόρφμαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ε, των προϊόντων που χρηματοδοτούμε. Το ευρωπαϊκό γάλα είναι πράσινο, λέμε. Παράδειγμα Ιταλία και Αυστρία. Μετά για τα κύβη Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία θα πρέπει να συμφωνήσουν για να εξαγάγουν κύβη, ακτινίδια και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα προγράμματα διαρκούν ένα με τρία χρόνια. Το απλό πρόγραμμα εκπροσωπεί μόνο μία χώρα. Το πολλαπλό πρόγραμμα εκπροσωπεί πολλές χώρες. Συμμετέχουν πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οργανώσεις. Ξέρω ότι ο Επίτροπος Χόγκαν θέλει να ασκήσει και οικονομική διπλωματία. Θα ταξιδέψει στο Μεξικό, Κολομβία, Κίνα και Ιαπωνία με Ευρωπαίους επιχειρηματίες για να προωθήσει τις εξαγωγές μας. Και Πού βρίσκεται το ψαχνό, στα χρήματα, αυτή είναι η κατανομή των κονδυλίων. Και μάλιστα μου συνέβη κάτι περίεργο. Συνήθω ε, στην Επιτροπή γίνεται περικοπή των κονδυλίων. Εμένα μου έδωσαν επιπλέον 30 εκατομμύρια, περισσότερο από πριν, χάρη στην κρίση στο χείριο και στο γαλακτοκομικό τομέα και τα βάλαμε στο 3 και στο 10. Ε, 9 συν 21 συγκεντρώνουμε τα 30 επιπλέον εκατομμύρια που έχουμε για τον τομέα χειρίου και το γαλακτοκομικό τομέα. Επίσης, πολλά κονδύλια τα διαθέσαμε σε τρίτες χώρες, ε, Ηνωμένε Πολιτείες, Κίνα. Αυτή είναι η κατανομή που γίνεται και είναι ενδεικτική η κατανομή. Την πρώτη χρονιά θα έχουμε 111 εκατομμύρια για να δαπανίσουμε σε πρόθεση των εξαγωγών μας, των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Και αυτό που θα ήθελα κύριε Πρόεδρε, και με αυτό θα ολοκληρώσω, θα ήθελα να με κατακλείσουν αιτήσει από όλη την Ευρώπη για να προωθήσουμε τις αγροεπιστηστικές μας εξαγωγές. Μακάρι να με βομβαρδίσουν με τέτοια αιτήματα, γιατί χρήματα υπάρχουν. Θα ήθελα λοιπόν ε, να διαδώσουμε τον, την καλή είδηση του νέου κανονισμού που μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ από τους γεωργούς και τις οργανώσεις. Παρακαλώ ε, θα ήθελα και εσείς να συμβάλλετε στην ε, περαιτέρω διάδοσή του γιατί είναι και δικό σας παιδί ο κανονισμός αυτός. Ευχαριστώ. Πρώτη ομιλητριά μας η κυρία Εράς Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Διέγκο Κάγκα για την παρουσίαση που μας έκανε του κανονισμού. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή και να δώσω τα εύσημα στον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, τον Επίτροπο τότε Τσόλος, ε, που μας βοήθησε πολύ και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα και με δύο μόνο τριμερείς διαλόγους καταλήξαμε σε συμφωνία τα τρία θεσμικά όργανα. Μετά την έγκριση του κανονισμού ανέκυψαν και ορισμένες μικρολεπτομέρειες και θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία της, για την προθυμία που έδειξε, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που ευτυχώς καταφέραμε και τις ε, διορθώσαμε. Ό,τι ζήτησε ο κλάδος ε, το καταφέραμε. Εγώ άκουσα εκπροσώπους στο γραφείο μου με προβληματισμό ε, για αναζήτηση εταίρων από άλλες περιοχές, ιδιαίτερα για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Μακάρι να ενισχυθούν τέτοιες συνεργασίες για να κάνουμε διαφοροποίηση των εξαγωγών και όταν συμβαίνουν τέτοιες κρίσεις όπως αυτή του ρωσικού εμπάργου να ξεφεύγουμε από την κρίση ανώδυνα για να μην πληρώνει πάντα πρωτογενής τομέας η γεωργία και η γεωργική παραγωγή τα σπασμένα τέτοιων κρίσεων. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και στον κύριο Χόγκαν που προωθεί το θέμα ως νέος επίτροπος. Του ευχόμαστε καλή τύχη στις εκστρατείες που θα κάνει στις τρίτες χώρες και επίσης ε, σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε την προσπάθεια για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονομασίες προέλευσης ε, να στείλετε μηνύματα σε όλες τις καταγεγραμμένες γεωγραφικές ενδείξεις για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα εκατομμύρια που έχετε στη διάθεσή σας για την πρόθεση των προϊόντων που θα συμβάλλει στη δημιουργία απασχόλησης ε, και στην καλύτερη πρόθεση των γεωργικών μας προϊόντων. Σας ευχαριστώ, κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ νομίζω ότι πρόκειται για καλές ειδήσει για την γεωργία στην Ευρώπη και πράγματι όπως εξελίσσονται οι αγορές πρέπει και εμείς να φανούμε επιθετικότεροι και να προωθήσουμε τα προϊόντα μας με ενισχυμένο τρόπο για να επιδείχουμε και καλύτερες τιμές. Κάτι που με ενδιαφέρει πολύ, το είπε και ο κύριος Γκραναφάνο, είναι ότι συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία αυτή και οι διάφορες ε, ε, διαβεβαιώσεις ποιότητας. Και χαίρομαι που προτείνει και μια ειδική ετικέτα γάλα από το βουνό. Στη φωτογραφία βέβαια δείχνει ένα ελβετικό βουνό και από ό,τι ξέρω η Ελβετία δεν είναι χώρα μέλος της Ένωσης. Αλλά τέλος πάντων αυτό μπορούμε και να το διορθώσουμε. Μέχρι τώρα πάντως η κατανομή των κονδυλίων αυτών ανάμεσα στην εσωτερική αγορά και, και στα προϊόντα που κατευθύνονται σε αγορές εκτός Ευρώπης. Πώς έχει γίνει μέχρι τώρα η κατανομή των κονδυλίων αυτών, πώς νομίζετε ότι εξελίσσεται. Και ποιο ποσοστό θα κατευθυνθεί σε υποστήριξη προγραμμάτων εξαγωγών εκτός Ευρώπης. Ευχαριστώ κυρία Γιλέρα. Σας ευχαριστώ. Όντως ε, πολύ καλή είδηση και μας δίνει και πολλές ευκαιρίες. Και όπως είπε ο κύριος Κάγκα, είχε ήδη κονδύλια και του έδωσαν περισσότερα, τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς. Θαυμάσια. Επίσης, να αποτίσω φορό τιμής στην κυρία Εράνς και στο σκιώδη δισηγητή, τον κύριο Γκαρσία, που ασχολήθηκα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό με το θέμα αυτό και χάρη σε όλη αυτή την προσπάθεια ευωδόθηκαν οι εργασίες μας. Κάποιες ερωτήσεις να κάνω τώρα. Ο κύριος Χόγκαν, ο Επίτροπος Χόγκαν, μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία διπλωμα... οικονομικής διπλωματίας ή διπλωματίας της οικονομίας στις εκστρατείες που θα κάνει. Μας αναφέρατε σε ποιες χώρες θα μεταβεί ο Επίτροπος. Ποιες επιχειρήσεις θα το, ποιοι επιχειρηματίες θα το συνοδεύουν, θα πρέπει να είναι επιχειρήσεις που ήδη έχουν υποβάλει αίτηση για συγχρηματοδότηση για την πρόθεση. Και Φαντάζομαι ότι ο Επίτροπος διάλεξε συγκεκριμένε αυτέ χώρε γιατί έχουν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την πρόθεση γιατί είναι καλύτερες αγορές για τα προϊόντα μας. Με τι κριτήρια γίνεται αυτή η επιλογή των χωρών για αυτή τη διπλωματική οικονομική αποστολή του Επιτρόπου. Ένα άλλο θέμα. Οι γεωγραφικές ενδείξεις ή ονομασίες προέλευσης ε, ήδη έχουν κονδύλια για την πρόθεσή τους με άλλα προγράμματα. Φαντάζομαι δεν θα είναι ασύμβατη χρηματοδότηση από τον τελευταίο κανονισμό και είναι σωρευτικά τα κονδύλια αυτά ή όχι. Γιατί Ήδη υπάρχουν κονδύλια προώθηση για τις γεωγραφικές ενδείξει και τις ονομασίες πρόέλευση από άλλα προγράμματα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει δυνατότητα παρόλα αυτά να υποβληθεί έτσι και με βάση τον τελευταίο κανονισμό. Ελπίζω να μην είναι ασύμβατο κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταντάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για αυτή την ανακοίνωση. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είδα ότι στην τελευταία διαφάνεια υπάρχουν κάποια στοιχεία επικοινωνίας αλλά με ποιο τρόπο θα μας ανακοινώνει τα, τις νέες πολιτικές η Κομισιόν ή αυτές τις ανασχεδιασμένες πολιτικές Βλέπουμε στα γραφικά ότι χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για τις πολιτικές εξαγωγών και μετά για τα προϊόντα ποιότητας και εδώ θα απαντήσω και για την προηγούμενη συζήτηση, θα, ε, θα για την προηγούμενη συζήτηση για τις επισημάνσεις για ορεινά προϊόντα. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι πολύ γνωστά μεταξύ καταναλωτών. Και επαναλαμβάνω κάτι που συχνά αναφέρουμε στην Επιτροπή Γεωργίας. Η Κομισιόν πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει μια ανακοίνωση μια εκστρατεία επικοινωνίας στο ευρύ κοινό για να ε, αναγνωρίζονται τα σήματα ποιότητας, ε, τα pop, ε, για τα ορεινά προϊόντα, γιατί όλα αυτά τα εργαλεία έχουν προκύψει μετά από πολλή δουλειά και προσθέτουν αξία, αλλά θα προσθέσουν αξία εφόσον είναι γνωστά στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στο κοινό των πόλεων, το οποίο δεν γνωρίζει αυτά τα σήματα ποιότητας. Ευχαριστώ. Κύριε Καγκοφάνο, έχετε και πάλι το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Eh, eh, eh. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Εράνς, γιατί εκείνη ήταν η συγγήτρια για τον κανονισμό. Χωρίς τη δική της παρουσία και συμβολή δεν θα είχαμε σήμερα κανονισμό, οπότε αμοιβέ είναι οι ευχαριστήσεις και τα συγχαρητήρια. Κύριε Ντόρφμαν, ε, η τάση ε, είναι περισσότερα κονδύλια προς την εξωτερική αγορά, όχι την εσωτερική. Και ε, μετά το ρωσικό εμπάργκο είχαμε εντυπωσιακή αλλαγή. Γιατί σήμερα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αρχίζουν τις διαφοροποίηση ακόμη και με λιγότερο γενναιόδορους κανόνες. Τώρα με περισσότερη γενναιοδορή και περισσότερους γενναιόδορους κανόνες φαντάζομαι θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εξαγωγών προς εξωτερικές αγορές. Γιατί δεν έχουμε μόνο τις παραδοσιακές αγορές Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Έχουμε και το Ντουμπάι, το Κατάρ, Αφρική, Λατινική Αμερική, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτή είναι η τάση προς εξωτερικές αγορές και ελπίζω να την ενισχύσει και ο νέος κανονισμός. Η οικονομική διπλωματία έχει έμεση σχέση με το θέμα αυτό ο Επίτροπο Χόγκα θα ξεκινήσει την επίσκεψη από το Μεξικό και την Κολοδία και μετά θα πάει στην Κίνα και την Ιαπωνία για να ανοίξει αγορέ. Ε, και μάλιστα ε, εθελοντές είναι οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που θα τον συνοδεύσουν. Ζητήσαμε εθελοντές ε, για το ταξίδι αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην αντιπροσωπεία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες. Πολλοί κόσμοι ενδιαφέρεται για να εκμεταλλευτεί αυτή την οικονομική διπλωματία που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την στήριξη που λαμβάνουν οι γεωρικές ενδείξεις και POP από άλλα προγράμματα. Καμία σχέση με τον κανονισμό. Εμεί θέλουμε να προωθήσουμε τις εξαγωγές με τον κανονισμό αυτό. Και έτσι θα αξιοποιηθούν τα κονδύλια. Οπότε δεν υπάρχει κανένα συμβίβαστο. Κύριε Νταντά, δίκιο έχετε ότι θέλουμε ο κανονισμό αυτό να ε, λάβει δημοσιότητα, να διαδοθεί, να εξαπλωθεί και αυτό εξαρτάται και από εσά, γιατί βρήθη ευκαιριών και δυνατοτήτων ο κανονισμός και καλό θα είναι να τον μάθει ο κόσμος. Ε, Εμεί ταξιδέψαμε στην Ευρώπη ε, και ο κύριος Χόγκαν ε, έκανε πολλές ανακοινώσεις, tweets στην ιστοσελίδα, αλλά δεν αρκεί. Βοηθήστε μας κι εσείς να μεταφέρουμε αυτή τη χαρμόσυνη είδηση του νέου κανονισμού. Και τέλος, για τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα. Υπάρχει και νομική υποχρέωση τα λογότυπα να μην είναι προαιρετικά, αλλά δεσμευτικά υποχρεωτικά και τα τρία λογότυπα του κανονισμού. Οπότε έτσι θα ε, γίνουν πιο γνωστά τα λογότυπα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι και πολύ γνωστά και κρίμα και έχουμε συμφέρον να γίνουν γνωστά τα λογότυπα όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο. Αυτά. Ευχαριστώ. porządek punktów merytorycznych. Bardzo dziękuję dobrze, że z taką nowiną Pan dzisiaj do nas przyszedł, że ten program wchodzi w życie.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 Θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε, στην δεξίωση, στον τρίτο όροφο, στις 6.30. Και είχα την αίσθηση ότι φέτος, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης ΚΑΠ, θα έχουμε λιγότερη δουλειά. Αλλά τελικά το αντίθετο έγινε. Είχαμε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Είχαμε τα ζωοτεχνικά θέματα, την έκθεση του κύριου Νταντά, το θέμα της κυρίας Αγγιλέρια, Επίσης είχαμε το ζήτημα της κλωνοποίησης, ε, θέμα με το οποίο είμαστε συναρμόδιοι με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρώτη φορά που είχαμε τέτοια συναρμοδιότητα δύο επιτροπών για την κλωνοποίηση. Επίσης σημαντική ήταν και η γνωμοδότηση της κυρίας Πάουλσεν. Πολύ σημαντική η συνεισφορά και αυτής της γνωμοδότησης. Επίσης είχαμε έκθεση για τη βιολογική γεωργία, πολύ σημαντικό θέμα και αρκετά επίμαχο. Γι' αυτό αρμόδιος είναι ο κύριος Χόισλινγκ. Επίσης ε, το ζήτημα της διανομής ε, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, θέμα του κυρίου Ταραμπέλα, θέματα γενετικής μηχανικής, ζήτημα που απασχόλησε την έκθεση της κυρίας Μακιντάιρ, επίσης ε, θέματα βελτιωση φυτών, την πολύ επικαιρή έκθεση του κυρίου Νίκολσον για την στρατηγική στο γαλακτοκομικό τομέα, γιατί γνωρίζουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στο γαλακτοκομικό κλάδο. Επίσης, ε, στρατηγική για τα δάση. Είχαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Θέματα επιστημικής ασφάλειας, δημοσιονομικά, εμπορικά, τη ΤΥΠ, ο κύριος Δεκάστρο, ο κύριος Νίκολσον ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά, μεταξύ άλλων. Μακροσκελής κατάλογος λοιπόν θεμάτων που θα συνεχιστεί και στο επόμενο έτος. Και μάλιστα η χρονιά αυτή ήταν δύσκολη για τους Γιώργους. Μεγάλες δυσκολίες προκλήθηκαν από το ρωσικό εμπάργο αλλά και η κατάργηση των γαλακτοκομικών προσωστώσεων δημιούργησε πρόβλημα. Φροντίσαμε όμως ε, να δώσουμε αποζημιώσεις, να στηρίξουμε τους γεωργούς για να αποφύγουμε την εμβάθυση της κρίσης. Και όπως ε, μας είπε και πρόσφυγος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπουμε την κόκκινη γραμμή ότι οι εξαγωγές μας ε, πάνε πολύ καλά. Σημαντικό αυτό. Βέβαια έχουμε πολλές προκλήσεις ακόμη μπροστά μας. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής, γιατί μέχρι στιγμή η συνεργασία μας ήταν πολύ αγαστή, παρόλο που το πρόγραμμά μας ήταν πολύ φορτωμένο, είχαμε και την έξπο του Μιλάνου. Μας ενημέρωσε γι' αυτό ο κύριος Δεκάστρο και δόθηκε ιδιαίτερη έφαση στη Γεωργία στην διεθνή αυτή έκθεση του Μιλάνου. Μερικές φορές δεν, συμφωνήσαμε, δεν συμφωνούσαμε, έχουμε διάσταση απόψεων, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ για να συζητάμε. Και από τη συζήτηση προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό ισχύει όχι μόνο στην Επιτροπή μας, γενικώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά και τη γραμματεία, τους συνεργάτες μας, τους βοηθούς μας. Χάρη στη δική σας ε, επίσης παρουσία και συνεργασία φτάνει το έργο της Επιτροπής και πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οργανώσεις, ε, στους παραγωγούς, σε όλους ε, όσοι ενδιαφέρονται για τα θέματα της γεωργίας. Αυτά ως προς τις ευχαριστίες. Σας εύχομαι καλές γιορτές, μια και είναι τελευταία συνεδρίαση πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και των νέο έτους. Μπορώ να ολοκληρώσω, έχουμε να προσθέσουμε τίποτα πριν περάσουμε στη Χριστουγεννιάτικη δεξίωση. Αμάν. Ξέχασα και την έκτακτη συνεδρίαση που έχουμε στις 9.30 την Πέμπτη, κοινή συνεδρίαση με τις Επιτροπές ΕΜΒΙ και ΝΤΕΒΕ, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Θα έχουμε μία ακόμη συνεδρίαση για τα εδάφη. Παρακαλώ δώστε το παρόν στην συνεδρίαση της Πέμπτης, ε, γιατί γίνεται επευκαιρία της ε, Διεθνούς ημέρας ε, για τα εδάφη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αναλάβει μέρος ε, στην συνεδρίαση αυτή και η Επιτροπή Γεωργίας, γιατί για μας τα εδάφη, οι είναι πολύ σημαντικές για τη Γεωργία. Πέμπτη λοιπόν, 9.30, μην ξεχάτε την κοινή αυτή, επιτροπή των την κοινή αυτή συνεδρία των τριών επιτροπών, Agri, Dev, Envy. Ευχαριστώ τη γραμματεία που μου το επενθύμησε. Αυτά πλησιάζουμε και την ώρα της δεξίωσης. Όπως είπα γίνεται στον τρίτο όροφο από τις 6.30 όσοι πιστοί προσέλθετε. Θα είναι μια σεμνή τελετή, μια δεξίωση εν ώψη των Χριστουγεννιάτικων διακοπών. Καλό σας βράδυ.